Well, good morning, everyone. Um, we are continuing our employment committee meeting left over from. Καλημέρα, θα συνεχίσουμε από εκεί που διακόψαμε εχθές. Θα ήθελα να σας πω ότι όλες οι γλώσσες εκτός από τα φιλανδικά, κροατικά, κελτικά και φιλανδικά είναι διαθέσιμα. Θα ήθελα επίσης να σας πω ότι λίγο αργότερα έχουμε και την ακρόαση για τους νέους. Νομίζω, νομίζω ότι περίπου 100 νέοι θα έρθουν. Και βεβαίως εδώ έχουμε μια πολύ μικρή αίθουσα. Συνήθως ε, δεν μπορούμε να ξεπεράσουμε τους 250 ε, και αν χρησιμοποιήσουμε όλες τις θέσεις όλων των ε, βοηθών, βουλευτών, αναπληρωτών. Φτάνουμε τους 190. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν να δούμε αν είναι δυνατόν να αφήσουμε κάποιες κενές θέσεις για τους νέους αυτούς, οι οποίοι ενδιαφέρονται να έρθουν και να ακούσουν αυτά τα οποία λέμε. Αν είναι δυνατόν δηλαδή να μαζευτούμε λίγο εδώ, για να τους αφήσουμε να καθίσουν και να συμμετάσχουν στο γεγονός αυτό. Ξεκινάμε όμως με τον Michael O'Flaherty, ο οποίος είναι ο Διευθυντής ε, της ε, Υπηρεσίας ε, Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Θα του δώσω 10 λεπτά περίπου το λόγο και κατόπιν θα δώσω το λόγο στον εκπρόσωπο του ILO, τον κύριο Εμμάνουελ Πόρ. Δεν υπάρχει κάποιος από την Επιτροπή παρόν στην αίθουσα. Κατόπιν λοιπόν θα δώσουμε το λόγο στα μέλη που θέλουν να συμμετάσχουν στη συζήτηση. Ο καθηγητής, ο κύριος Οφλάρτη, έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρος, διακεκριμένα μέλη της Επιτροπής, αγαπητοί φίλοι, εξ ονόματις ε, του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων θα ήθελα να σας πω ότι είναι μεγάλη τιμή για μένα που απευθύνομαι σε εσά. Θεωρούμε ότι το έργο τη Επιτροπής σα είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τα ανθρώπινα και θεμελιώδη δικαιώματα. Αναφερόμενο σε δύο παραδείγματα με επηρεάζει σημασία του άρθρου 15 της χάρτης που εξασφαλίζει στους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης το δικαίωμα να αναζητήσουν εργασία και να προσφέρουν εργασία σε οποιοδήποτε κράτος μέλος. Το άρθρο 31 που διασφαλίζει ε, το δικαίωμα σε δίκες και ίσες ε, συνθήκες εργασίας. Γι' αυτό το λόγο αισθάνομαι πολύ άνετα σήμερα μεταξύ σας. Να λάβετε υπόψη επίσης ότι τα δικαιώματα στην απασχόληση είναι να πολλαπλασιαστή για να μπορεί να απολαύσει κανείς πολλές άλλες ελευθερίες. Ε, κληθήκαμε να σας μιλήσουμε σήμερα το πρωί για τους τομείς ε, της εργασίας μας που επικαλύπτονται με τον τομέα των αρμοδιοτήτων σας κυρίως όσον αφορά τις σοβαρές μορφές εκμετάλλευσης εργασίας. Θα έλθω σε αυτό το θέμα αμέσως. Όταν μιλάμε για σοβαρή εκμετάλλευση στην εργασία, αναφερόμαστε στις μορφές εκμετάλλευση εργασίας που είναι είτε εγκληματικές, σύμφωνα με την νομοθεσία των κρατών μελών, ή μπορούν να ποινικοποιηθούν σύμφωνα με ε, το διεθνή ή ενωσιακό νόμο. Περιλαμβάνονται πρακτικές όπως η δουλεία, η εξαναγκαστική εργασία, όλες οι, οι μορφές εκμετάλλευσης που πρέπει να απεικονοποιηθούν στα πλαίσια της οδηγίας επιβολής ποινή ε, στους εργοδότες. Μεταξύ του 2013 και 2015 ο οργανισμό μας έκανε μεγάλες έρευνες στα φαινόμενα αυτής της ε, εκμετάλλευση των εργαζομένων σε όλα τα κράτη-μέλη. Και το αποτέλεσμα η έκθεση, ήταν μια έκθεση η οποία ξεκίνησε το 2015, είναι η μόνη έκθεση αυτής της μορφής που εξετάζει ε, όλες τις μορφές εκμετάλλευση στην εργασία. Παρουσιάζει τις απόψεις 600 επαγγελματιών σε 21 κράτη-μέλη και όσον αφορά τους τομείς που συμβάλλουν στην εκμετάλλευση, ε, επίσης ε, προτείνει τρόπους για την πρόθεση ε, πρακτικών που υπόσχονται πολλά. Ανάμεσα ε, στα βασικά πορίσματα αυτής της εργασίας του οργανισμού μας αναφέρουμε ότι υπάρχει μεγάλη συχνότητα σοβαρής εκμετάλλευσης στην εργασία. Αλλά οι υπεύθυνοι σπανίως διώκονται ή καταδικάζονται. Κατά κάποιο τρόπο αυτό είναι ανησυχητικό σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση όπου υπάρχει αυτό το σύστημα ατιμορρησίας που βασίζεται σε τρεις πυλώνες. Ο πρώτος είναι κατακαιρματισμός των διατάξεων του ποινικού, δεύτερον έλλειψη παρακολούθησης και τρίτον η έλλειψη προληπτικών πολιτικών και πρωτοβουλειών και ερευνών. Επίσης η έρευνά μας επισημαίνει ότι αυτές οι μορφές εκμετάλλευση στην εργασία υπάρχουν σε ορισμένους τομείς, τη γεωργία, ε, τις κατασκευές, τη στέγαση ε, και τις υπηρεσίες εστίασης και τέλος ε, στις οικιακές εργασίες. Με χαρά ενημερώνω την Επιτροπή ότι με βάση αυτή την έκθεση ο οργανισμός μας εξακολούθησε τις έρευνες του σε αυτόν τον τομέα και το 1917 θα παρουσιάσει μια νέα έκθεση που θα καλύπτει τις απόψεις των αλλοδαπών εργαζομένων. Με αυτόν τον τρόπο η έρευνα ε, θα πληρώσει ένα σημαντικό κενό ε, δεδομένου ότι όχι μόνο θα εξηγήσει τι συμβαίνει από την πλευρά των επαγγελματιών, αλλά και από την πλευρά εκείνων που πλήττονται περισσότερο, δηλαδή οι ίδιοι εργαζόμενοι. Πιστεύουμε λοιπόν ότι ως αποτέλεσμα η νέα έρευνα του 2017 με βάση τα αποτελέσματα του 2015 θα οδηγήσουν σε σημαντικά μέτρα υποστήριξης για σας προκειμένου να διαμορφωθούν σωστές πολιτικές και νομοθεσίες. Πριν λοιπόν από τα πορίσματα του 2017, θα ήθελα με κάθε σεβασμό να σας προτείνω οι συστάσεις που κάναμε το 2015 να παραμείνουν έγκυρες και να λυθούν υπόψη. Μεταξύ αυτών τονίζουμε τις εξή. Πρώτον, η ανάγκη να δημιουργηθούν, να δημιουργηθούν ορισμοί κατανοητοί που προστατεύουν όλους τους εργαζόμενους κατά της σοβαρής εκμετάλλευσης. Δεύτερον, η μεγαλύτερη παρακολούθηση από επιθεωρήσεις εργασία από τα συνδικάτα, από την ε, αστυνομία του οικονομικού εγκλήματος που έχουν επαρκείς πόρους και αρμοδιότητα για να φέρουν εις πέρα στο έργο τους. Τρίτον, η ανάγκη να δημιουργηθούν συστήματα ε, κυκού branding που είναι αξιόπιστα και που επιτρέπουν στους καταναλωτές να γνωρίζουν πότε υπάρχει ε, κίνδυνος ε, εκμετάλλευσης. Τέλος, να εξασφαλίσουμε ότι οι πολίτες της Ευρώπης που αποφασίζουν να δουλέψουν σε ένα άλλο κράτος μέλος ενημερώνονται εκ των προτέρων για τους κινδύνους εκμετάλλευσης και πού μπορούν να στραφούν αν χρειάζονται βοήθεια. Νομίζω το θέμα ε, των σοβαρών μορφών εκμετάλλευσης εργασίας είναι πολύ σημαντικό και θα ήθελα τώρα να θίξω δύο άλλου τομεί όπου δραστηριοποιούμεθα και παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την εργασία τη επιτροπή. Πρώτα απ' όλα η κατάσταση των Ρωμά. Οι Ρωμά, όπως γνωρίζετε, είναι η μεγαλύτερη μειονότητα στην Ευρώπη, εκείνη που πλήττεται περισσότερο από διακρίσεις η προηγούμενη εργασία του οργανισμού μας ε, δείχνει ότι αντιμετωπίζουν πολλές δυσκολίες οι Ρωμά στις εργασιακές τους σχέσεις. Χαμηλές αμοιβέ, κυρίως για τους νέους Ρωμά, έλλειψη ε, προσόντων, παιδείας, σε συνδυασμό με ε, μια διάκριση. Όλα αυτά ενισχύουν τον αποκλεισμό τους από την επίσημη αγορά εργασίας. Ο οργανισμός μας θα δημοσιεύσει νέα στοιχεία στο τέλος του μηνός, 28 Νοεμβρίου, για τους Ρωμά. Και λυπούμε να σας αναφέρω ότι τα αποτελέσματα αυτά είναι ανησυχητικά. Μεταξύ ε, των ε, αποτελεσμάτων που θα δημοσιευθούν σε δύο εβδομάδε δείχνουν ότι 20% μόνο των Ρωμά μεταξύ 20 και 68 ετών αμείβονται ε, στη δουλειά τους. Δηλαδή, αυτό είναι ένα μεγάλο ποσοστό. Ε, όσον αφορά τους νέους, μόνο 37% των νέων Ρωμά ε, απασχολούνται, εκπαιδεύονται ή επιμορφώνονται. Αυτά είναι ανησυχητικά στοιχεία. Και μεταξύ άλλων δείχνουν ότι είναι για να επιτύχουμε ε, τον στόχο της σύστασης του Συμβουλίου του 2013 να λάβουμε αποτελεσματικά μέτρα για ίση μεταχείριση των Ρώμα και πρόοδο στην αγορά εργασία και στις ευκαιρίες απασχόλησης θα είναι ένα μεγάλο πρόβλημα όσον αφορά την εφαρμογή αυτής της οδηγία. Τέλος, αξιότιμα μέλη, θα ήθελα να μιλήσω για τα θέματα της έλλειψης ικανότητας των αναπηριών. Αναγνωρίζεται από τη χάρτα ε, τα δικαιώματα των ατόμων που έχουν αναπηρία να εργάζονται ίσης όρις με άλλους. Η Επιτροπή είναι μία από τις τρεις επιτροπές του Κοινοβουλίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια της Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Ανθρώπων με Αναπηρία και γνωρίζετε πολύ καλά τα θέματα τα οποία διακυβεύονται. Ο οργανισμός μας, επίσης, έχει καταλήξει σε στοιχεία απογοητευτικά. Οι τελευταίες στατιστικές από τη Συνδική Υπηρεσία ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ε, τα εισοδήματα και τις συνθήκες εργασίας του 2013 δείχνουν ότι υπάρχει μία απόκληση κατά 23% ε, των σχέσεων σε σχέση Δηλαδή, 23% απασχολούνται άτομα ανάπηρα σε σχέση με 70% χωρίς αναπηρία. Πρέπει να καλύψουν αυτό το κενό. Και γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να εφαρμοστούν ορισμένες πρακτικές στα κράτη-μέλη, δηλαδή και κίνητρα και ποσοστώσεις που είναι σημαντικές πρωτοβουλίες. Τα κίνητρα στην Πορτογαλία, για παράδειγμα, η Πορτογαλία παρέχει πολλά κονδύλια σε δημόσιους οργανισμούς για να προσλάβουν γυναίκες με αναπηρία ε, προκειμένου να προσληφθούν ή να ε, καταρτιστούν οι ο νόμος τη Κροατία για την επαγγελματική αποκατάσταση και την απασχόληση των ανθρώπων με αναπηρία αναγκάζει ε, τους εργοδότες να απασχολήσουν 20 άτομα ε, με αναπηρία. Αυτά είναι παραδείγματα ενδεικτικά των θετικών πρωτοβουλειών που βρίσκουμε στα κράτη-μέλη και που θα πρέπει να εφαρμοστούν και από άλλα κράτη-μέλη για να καταβάλουμε σημαντική προσπάθεια και να καλύψουμε αυτό το κενό το οποίο είναι απαράδεκτο. Κυρία Πρόεδρε, θα σταματήσω εδώ. Ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων είναι στη διάθεσή σας σήμερα το πρωί για τυχόν ερωτήματα που θα προκύψουν από τα μέλη της Επιτροπής. Υπάρχει ο Άλμπερ Ντίρινγκ ε, που είναι έμπειρος συνάδελφος και θέλει να σας εξασφαλίσω ότι ο οργανισμός μας εξακολουθεί να είναι στην υπηρεσία σας για να σας υποστηρίξει στο σημαντικό έργο που επιτελείτε. Ευχαριστώ πολύ. Now we'll invite... Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Εμάιν Πορ έχει το λόγο για πέντε λεπτά. Ευχαριστώ. Καλημέρα σε όλους. Είναι μεγάλη χαρά για μένα που μπορώ να πάρω το λόγο εδώ σήμερα το πρωί. Θα κάνω βεβαίως μια πρώτη παρουσίαση, κατόπιν θα είμαι στη διάθεσή σας ε, για την απάντηση τυχόν ερωτήσεων. Στην πράξη θα έπρεπε να γνωρίζετε ότι η κατάσταση είναι εξαιρετικά δύσκολη. Ακούσατε ήδη μία πρώτη παρουσίαση αλλά σήμερα έχουμε τουλάχιστον ένα εκατομμύριο άτομα τα οποία εργάζονται σε καταναγκαστική εργασία, 22 εκατομμύρια με άθλιες συνθήκες και εάν συγκρίνουμε αυτά τα 21 εκατομμύρια που είναι θύματα εκμετάλλευσης με τις 6.000 που έχουν προσφύγει στα δικαστήρια, καταλαβαίνετε ότι ε, τα πράγματα δεν είναι καθόλου απλά. Πολύ πρόσφατα το ILO έχει ήδη ασχοληθεί με όλες αυτές τις υποθέσεις, τις υποθέσεις και όλες τις υποθέσεις εκμετάλλευσης παιδιών, γυναικών και άθλιες συνθήκες εργασίας. Σκοπός μας είναι να φτάσουμε τον, τείχο, τον στόχο 8,7 8,7 και σας καλώ όλους να μπορέσετε να έχετε πρόσβαση στα στοιχεία που διαθέτουμε και να μπορέσετε να πληροφορηθείτε για όλες αυτές τις ε, υποθέσεις. Το πρωτόκολλο για την καταναγκαστική εργασία που πριν από δύο χρόνια προέκυψε από την ε, συνάντηση που είχαμε, που, οργανώσαμε στον ΑΕΛΟ και σας ε, προσκαλώ όλους να κοιτάξετε το θέμα της κύρωσης αυτού του πρωτοκόλλου. Είναι κάτι που Πιστεύω ότι το οφείλουμε τουλάχιστον σε όλους αυτούς τα 21 εκατομμύρια θύματα της ε, εκμετάλλευσης της καταναγκαστικής εργασίας. Μιλάμε για 150 δισεκατομμύρια δολάρια. Είναι το ποσό των κερδών που προκύπτουν από αυτό το τομέα της καταναγκαστικής εργασίας. Πρόκειται για ένα τεράστιο ποσό και αν θέλουμε να το εξαλείψουμε Φυσικά και θα πρέπει να καταπολεμήσουμε τις ρίζες αυτού του φαινομένου. Καταλαβαίνετε ότι η δράση μας είναι ε, κάτι που θα πρέπει να μας απασχολήσει όλοι και είναι επίγον το θέμα αυτό. Είμαι στη διάθεσή σας για απάντηση τυχόν ερωτήσεων. Πρόεδρος. Όποιος ε, θα ήθελε να πάρει το λόγο, βλέπω την Χέλγα Στίβενς από την ECR, την κυρία Κάρη, δεν ξέρω ποιος άλλος θα ήθελε να πάρει το λόγο. Ξεκινάμε με την Χάλικα Στίβενς. Uh, uh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε, και μέσα στην αδελφή. Ευχαριστώ για τα θέματα που αναφέρατε και θα ήθελα να αφαιρθώ στους εργαζόμενους με αναπηρία. Πρώτα να πω όμως ότι για τις καταχρήσεις φαίνεται να έχουμε μια μετατόπιση προς οργανωμένες εγκληματικές δραστηριότητες σε σχέση με την παρουσία συμμοριών που παρεσφρίουν σε χώρους εργασίας για να εκμεταλλευτούν ακριβώς εργαζομένους. Πολλές χώρες μέλη έχουν λάβει ενεργά μέτρα για να αντιμετωπίσουν την παράνομη εργασία σε όλους τους κλάδους. Παρ' αυτά Χρειάζεται περισσότερη ηγεσία και μεγαλύτερε προσπάθειες μεταξύ των διαφόρων αρχών των χωρών μελών για να έχουμε μια πιο στοχευμένη δράση ώστε να σταματήσουμε την εκμετάλλευση, να πετύχουμε τη συμμόρφωση και να επιφέρουμε επίση και κάποια ευελιξία όσον αφορά την συμμόρφωση σε εθνικό επίπεδο. Επίση, θα πρέπει να θυμόμαστε ότι η εκμετάλλευση είναι κάτω διεθνέ, οπότε απαιτεί διεθνή αντίδραση. Αντί λοιπόν κάθε χώρα να κυνηγά μόνη της στο εσωτερικό της εγκληματίες, όπως αναφέρθηκε, ίσως να χρειαζόμαστε μια νέα συνολική προσέγγιση για να καθορίσουμε αυτό το νέο επιχειρηματικό μοντέλο και να το αντιμετωπίσουμε, ώστε να διασφαλίσουμε και ότι η Ευρώπη και τα μέλη της θα συνεργαστούν με τους διεθνείς εταίρους με τρόπο αποτελεσματικό. Έχω λοιπόν κάποιες ερωτήσεις να υποβάλω. Στην έρευνα σας είδατε μήπως κάποια αύξηση της εκμετάλλευσης τα τελευταία χρόνια σε κάποιο συγκεκριμένο κλάδο ή σε κάποιο τομέα της κοινωνίας ή μήπως αυτή η εκμετάλλευση αφορά υπηκόους τρίτων χωρών ή υπηκόους χωρών της Ένωσης. Έχετε επίσης παραδείγματα καλών πρακτικών για τα μέτρα που λαμβάνουν τα ενεργά οι χώρε μέλη για να καταπολεμήσουν την εκμετάλλευση. Α πούμε, στο Ηνωμένο Βασίλειο υπάρχει ο νόμο για τη σύγχρονη σκλαβιά που θεσπίστηκε το 2015, πρώτο νόμο αυτού του είδου στην Ένωση. Η Ένωση λοιπόν πώ θα μπορούσε να συνεργαστεί με τι χώρε μέλη για αυτά τα θέματα, α πούμε, μέσω τη ανταλλαγή πληροφοριών. Και να μιλήσω τώρα για τα άτομα με αναπηρία και την απασχόληση. Είπατε ότι είχαμε κάποια ποσοστά χαμηλότερα σε σχέση αυτό που έχουν αναπτύξει, σε σχέση με τα υψηλότερα αυτό που δεν έχουν. Μήπως εδώ ως πιθανή λύση θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι το οποίο θα έπρεπε να εστιάζεται σε στόχους και όχι τόσο σε ποσοστά. Μήπως θα έπρεπε να δούμε τι υπάρχει ή τι βρίσκεται πίσω από τα ποσοστά. Γιατί λένε πολλές επιχειρήσεις ότι εμείς τηρούμε τις υποχρεώσεις μας, όμως θα πρέπει να δείτε πού δουλεύουν αυτά τα άτομα με αναπηρία στο εσωτερικό της επιχείρησης. Ας πούμε, προσλαμβάνουν καθαριστές και για να τηρήσουν τις ποσοστώσεις τους. Έχουν όμως αυτά τα άτομα ευκαιρίες ε, ανέλυξης, ευκαιρίες κατάρτισης κλπ. Θα ήθελα λοιπόν να μου πείτε εδώ τι γίνεται. Επίσης υπάρχει ένα θέμα με το επίπεδο εκπαίδευσης. Συχνά αυτά τα άτομα με αναπηρίες δεν έχουν τις ίδιες ευκαιρίες εκπαίδευσης όπως τα άτομα χωρίς αναπηρία. Αυτό λοιπόν έχει επιπτώσεις όσον αφορά τις ευκαιρίες τους στην αγορά εργασίας. Όπως λέγαμε λοιπόν, θα πρέπει να ξεκινήσουμε με υψηλά πρότυπα Εκπαίδευση για τα άτομα και για τα παιδιά με αναπηρία. Αυτό νομίζω είναι από τα βασικότερα με την βασική εκπαίδευση και μετά θα δούμε τι γίνεται με την εκπαίδευση που χρειάζεται για την έβρεση εργασία. Επίση, θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με την επιβολή για τι ποσοστώσει. Είδαμε μελέτε στη Γαλλία και στη Γερμανία που δείχνουν ότι οι επιχειρήσει δεν προτιμούν να προσλαμβάνουν άτομα με αναπηρία, ε, προτιμούν να πληρώσουν το πρόστιμο, όποιο και αν είναι αυτό. Οπότε, μήπως εδώ πρέπει να αλλάξουμε τη στάση αυτή και να προωθήσουμε την ένταξη και την περίληψη των ατόμων με αναπηρία στην αγορά εργασία, Να έχουμε δηλαδή περιεκτική απασχόληση μαζί με την αντίστοιχη εκπαίδευση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Έχω πέντε ομιλητέ. Θα του ακούσουμε και θα απαντήσουν μετά οι ομιλητέ μα. Γκουερίνα Καρή. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα μιλήσω δανεικά. Καταρχάς, σας ευχαριστώ και τους δύο για αυτά τα αρχικά σχόλια. Όντως, το θέμα αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό. Το έχουμε συζητήσει επανειλημμένως εδώ στην Επιτροπή μας και το παίρνουμε πολύ σοβαρά. Δύο ερωτήσεις έχω. Πρώτη ερώτηση. Όταν μιλάμε για συστάσεις, για το γεγονό δηλαδή ότι θα πρέπει να γίνουν περισσότερα σε επίπεδο επιθεωρητών εργασία, συνδικάτων κτλ. Μπορείτε να είστε πιο συγκεκριμένοι. Τι μπορεί να γίνει πιο αποτελεσματικά. Στη Δανία, α πούμε, είδαμε ότι είχαμε μεγαλύτερη εμπλοκή, μεγαλύτερη συμμετοχή των εργοδοτών μετά από κάποιες δικές μας αντιδράσεις. Μετά όμως μετατόπισαν τις θέσεις εργασία οι εργοδότες με τον ίδιο βαθμό εκμετάλλευσης. Οπότε τι μπορούμε να κάνουμε ώστε να μην υπάρχει τρόπος αποφυγής των ελέγχων. Μετά, για τα πρωτόκολλα του Διεθνούς ε, Διεθνής Οργάνωσης Εργασίας. Τι γίνεται εδώ, μπορείτε να μας πείτε τι γίνεται με αυτά τα πρωτόκολλα. Θα ήθελα να μας το πείτε ναι, για να δούμε ακριβώ, κατά πόσο θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε σύμφωνα με αυτά τα πρωτόκολλα που έχει στη διάθεση του Εθνικού Οργανισμού Εργασίας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ντομινίκ ε, Μαρτά, ΙΕΝΕΦ. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Ευχαριστώ ιδιαίτερος τον κύριο Φλάκετη για τα στοιχεία που μας ανέφερε. Το τι χρειάζεται να αποδείξουμε δηλαδή. Το είπατε κι εσείς. Αυτό που λέμε εμείς εδώ και χρόνια. Τα πρώτα θύματα δηλαδή της μετανάστευσης είναι ακριβώς οι ίδιοι μετανάστες. Το είπατε ξεκάθαρα εσείς ότι είναι αντικείμενο εκμετάλλευσης παρά τη θέλησή τους στην οικοδομή, στη γεωργία ή στην κατοίκο απασχόληση. Αυτή στην κατοικο αυτη η διαπιστωση σας λοιπόν με χαροποιεί. Αντίστροφα. Δηλαδή, τα πρώτα θύματα είναι μετανάστες. Οπότε οι μετανάστες δεν θα πρέπει να δέχονται επιθέσεις. Θα πρέπει λοιπόν αν χρειάζεται να κάνουμε κάτι τέτοιο, να επιτεθούμε στην μετανάστευση. Κατά συνέπεια ρωτάω και προτείνω ταυτόχρονα. Νομίζω ότι ο καλύτερος τρόπος για να προστατεύσουμε τους ξένους εργάτες είναι καταρχάς να αλλάξουμε τα σύνορα, τα σύνορα τους, αυτό δεν το αναφέραμε. Αυτός ο κόσμος δεν έρχεται εδώ στην τύχη. Μετά να ρυθμίσουμε τη μεταναστευτική ροή εσείς αυτό δεν το αναφέρατε. Βεβαίως οι ξένοι εργάτες έχουν τεχνογνωσία στο μέτρο όπου το χρειαζόμαστε αυτό. Αν δεν το χρειαζόμαστε δεν έχουν μέλλον. Αυτό το λέμε ρύθμιση. Τρίτον, θα πρέπει να κάνουμε κάτι με τους διακινητές, γιατί αυτοί έρχονται μόνοι τους οι διακινητές λοιπόν τους υπόσχονται ότι θα βρουν τον ε, παράδεισο. Τους λένε ψέματα. Το Ελντοράντο υπόσχονται σε αυτούς τους ξένους. Το οποίο όμως δεν ισχύει. Ακούσαμε προηγουμένως και για την σεξουαλική εκμετάλλευση αυτών των ξένων εργαζομένων. Θα πρέπει λοιπόν να αντιμετωπίσουμε αυτούς τους διακινητές που υπόσχονται ψέματα με αντάλλαγμα βέβαια υψηλά χρηματικά ποσά. Βεβαίω υπάρχουν επιχειρήσει οι οποίε εκμεταλλεύονται του ξένου εργαζομένου, θα πρέπει να τιμωρούνται, να τιμωρούνται. Υπάρχουν όμω επίση και συστήματα διακινητών με εκατομμύρια ευρώ που εκμεταλλεύονται αυτά τα άτομα. Οπότε χαίρομαι κύριε που σας άκουσα. Αυτά είχα να πω. Ευχαριστώ. Thank you. And our next speaker is Mr. Lopez for S&D. Muchísimas gracias, <clears throat> Presidenta. Yo tengo dos preguntas. A... Ευχαριστώ. Έχω δύο ερωτήσεις προς τους συζητητές. Καταρχάς για την εκμετάλλευση στην εργασία που αφορά τους μετανάστες, όπως είπατε. Να ρωτήσω όμως θεωρείτε ότι μεταρρυθμίσεις στον τομέα τη εργασία, όπως είχαμε τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα αυτές που έχουν εξασθενήσει τις συλλογικέ συμβάσει, αυτά είχαν επιπτώσει ενδεχομένω στα, στα θεμελιώδη δικαιώματα που έχουν οι πολίτε ιδιαίτερα στην αγορά εργασία και στη συμμετοχή του εκεί. Γιατί όπω ξέρουμε πολύ καλά είχαμε ε, μεταρρυθμίσεις ε, πολύ επιθετικές, οι αλλαγές είναι πολύ βαθιές αφορούν την εποχικότητα, νέο είδο συμβάσεων κλπ. Και κατά πόσο και αυτό το τελευταίο συνδέεται με την απώλεια βασικών δικαιωμάτων. Δεύτερη ερώτηση, όχι τόσο για την εκμετάλλευση, όπως είπατε εσείς, αλλά για τα οικονομικά και κοινωνικά δικαιώματα των πολιτών. Θεωρείτε ότι στην εργασία αυτή τη στιγμή που κάνει το Κοινοβούλιο και η Κομισιόν για την ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Πυλώνα. Θα μπορούσε η Ένωση λοιπόν να προωθήσει ένα θεματολόγιο οικονομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων. Η τελευταία δηλαδή γενιά δικαιωμάτων που θα πρέπει να προστατεύσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Και τελευταία ομιλήτρια είναι η κυρία Ευχαριστώ κύριε, κυρία Πρόεδρε. Ορισμένες συμπληρωματικές παρατηρήσεις. Δεν μιλήσατε για την διάκριση σε βάρος των γυναικών. Τη στιγμή όπου σε πολλές χώρες Ευρώπης επισύρουν την προσοχή γυναίκες για τη διαφορά των μισθών, αυτή η διάκριση θα πρέπει να υπογραμμιστεί, διότι συμβαίνει σε εμά, στην Ευρώπη, στις χώρες που υποτίθεται ότι είναι αναπτυγμένες και πιο προηγμένες σε σχέση με τον υπόλοιπο κόσμο. Ένα άλλο στοιχείο σχετικά με τη διάκριση στην εργασία είναι η κατηγορία των λεγόμενων ηλικιωμένων ατόμων. Στην Ευρώπη γυράσει κανείς όλο και πιο νέος, δηλαδή αποκλείεται από την αγορά εργασίας πολύ πιο νωρίς, επειδή σήμερα το κριτήριο της επιλογής είναι να έχει κανείς μεταξύ 20 και 30 χρονών και μετά τα 40 ήδη θεωρείται μεγάλη ηλικία για να προσληφθεί. Λοιπόν, αν μια επαγγελματική κατηγορία ε, η οποία δέχεται διάκριση είναι αυτή, το μεγαλύτερη ηλικία ατόμων. Επίσης υπογραμμίσατε την ανάγκη, ε, την υποχρέωση του ρόλου και το ρόλο των συνδικαλιστικών οργανώσεων. Και αυτό συμβαίνει στην Ευρώπη. Όλο και περισσότερο η συνδικαλιστική δράση ποινικοποιείται. Όλο και πιο πολλές προσφυγές στη δικαιοσύνη υπάρχουν κατά των συνδικάτων και της συνδικαλιστικής δράσης. Το υπογράμμισα και εσείς υπογραμμίσατε την σημασία της παρουσίας των συνδικάτων στις επιχειρήσεις όπου υπάρχει συνδικαλιστική παρουσία. Αυτό βλέπουμε ότι δεν υπάρχει τόσο μεγάλη διάκριση κατά των γυναικών, των μεγαλύτερης ηλικίας ατόμων, των αναπηρών ατόμων, των, των εργαζομένων και το καθεξής. Και υπάρχει, υπάρχουν μηχανισμοί, εργαλεία τα οποία μπορούν να καταστούν σχεδόν υποχρεωτικά. Και υπάρχουν σε ορισμένε χώρε, δηλαδή υποχρέωση να δημοσιοποιηθεί μια ετήσια έκθεση για του ανθρώπινου πόρου, για την παρουσία των εργαζομένων σε μια επιχείρηση. Και να γίνεται διάκριση μεταξύ των συνδικών εργασία, των θέσεων εργασία, των μισθών κ.ο.κ ποιος δουλεύει σε εμά. Αυτό δείχνει διαφάνεια και θα μπορούσε να είναι ένα εργαλείο πολύ σημαντικό για την καταπολέμηση όλων των διακρίσεων, κυρίως ε, της εξαναγκαστικής εργασίας, ε, της οποίας είναι θύματα πολύ συμπολίτε μας συμπεριλαμβανομένων των μεταναστών. Ευχαριστώ. Thank you. Ευχαριστώ. Επανέρχομαι στους δύο καλεσμένους μας και δίνω το ρόλο πρώτα στον κύριο Χάτερη. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα απαντήσω σε ορισμένα από τα ερωτήματα και ο συνάδελφός μου ο κύριος Deering θα δώσει τις πιο τεχνικές ερωτήσεις. Πρώτα απ' όλα, όσον αφορά το, το, τα ενδιαφέροντα ερωτήματα τη κυρία Ήβαν, θα ήθελα να παρακαλέσω τον κύριο Ντίερινγκ να απαντήσει στο θέμα των ε, ε, ακραίων μορφών εργασίας. Και εγώ θα μιλήσω για τα θέματα αναπηρίας. Συμφωνώ ότι είναι σκληρές οι ποσοστώσεις. Δεν είναι καθόλου μια ιδανική κατάσταση. Είναι μια ειλικρινή προσπάθεια να αντιμετωπίσει κανείς μια παράδεικτη κατάσταση. Η προσπάθεια αυτή είναι δύσκολη και συμφωνώ ότι πρέπει να παρακολουθούνται προσεκτικά και πρέπει να δει πίσω από τι ποσοστώσει την ποιότητα τη παρεχόμενη εργασία. Συμφωνώ λοιπόν ότι πράγματι είναι ένα τομέα που θα πρέπει να προσελκύσει την προσοχή μας. Συμφωνώ επίσης ότι η πρόσβαση στην παιδεία και στην εργασία είναι ένα σημαντικό θέμα, όχι μόνο όσον αφορά τα άτομα με αναπηρία, το ίδιο θα έλεγα για τους Ρωμά, για παράδειγμα. Αλλά δεν πρέπει κανείς να παραβλέπει τη σχέση ανάμεσα στην καλή παιδεία και τη σωστή δουλειά, την αξιοπρεπή δουλειά. Επίσης, απαντώντας ε, στην κυρία θα ήθελα να μιλήσω για το θέμα της ε, εφαρμογής και επίσης όταν υπάρχει η εκμετάλλευση. Ε, είπα ότι δεν υπάρχει αποτελεσματική εφαρμογή των μέτρων σε όλα τα κράτη-μέλη. Τώρα, για τα ερωτήματα, η κυρία Κάρη μίλησε για το θέμα της εφαρμογής, μιλήσατε για την παρακολούθηση και πώς γίνεται παρακολούθηση, παρατήρηση και μετά βρίσκουν νέα τεχνάσματα για να εκμεταλλευτούν τους εργαζόμενους. Όταν πρέπει να πούμε ότι υπάρχει πάντοτε η έλλειψη της πραγματικής βούλησης σε πολλά κράτη-μέλη να αντιμετωπίσουν αυτό το πρόβλημα. Ποιοι είναι τα θύματα των ακραίων μορφών εκμετάλλευσης στην εργασία. Δεν είναι τα άτομα που βρίσκονται στις ομάδες, στις κεντρικές ομάδες, αλλά στην περιφέρεια της κοινωνίας και αυτά στο περιθώριο της κοινωνίας. Και αυτά τα άτομα δεν τα λαμβάνουμε υπόψη όταν χαράζουμε τις πολιτικές. Ε, κύριε Μακάπ, μιλήσατε για το θέμα ε, των συνόρων. Απαντώντας την παρατηρήσή σας, θα ήθελα να πω ότι η μελέτη μας ασχολήθηκε με την μετανάστευση γενικά. Συμπεριλαμβάνονται και οι εξωευρωπαϊκοί. Γι' αυτό υπάρχει βεβαίω και μετανάστευση μεταξύ κρατών μελών της Ευρώπης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εκτός. Όσον αφορά τους αλλοδαπούς αφιχθέντες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κάναμε μελέτη για να δούμε ε, σε σχέση με την κρίση της μετανάστευσης και εντυπωσιαστήκαμε σε ποιο βαθμό τα άτομα που έρχονται στην Ευρώπη δεν είναι οικονομικοί μετανάστες, ε, αλλά προσπαθούν να διαφύγουν από τις διώξεις. Και το 2015, στα πλαίσια της κρίσης, τα περισσότερα άτομα έρχονται από τις ε, μεγαλύτερες χώρες από τις οποίες φεύγουν οι πρόσφυγες. Κύριε Λούκας, ζητήσατε σε ποιο βαθμό η εργατική νομοθεσία και οι συλλογικές διαπραγματεύσεις μπορούν να κάνουν διαφορά. Μπορεί ο συνάδελφός μας να απαντήσει σε περισσότερες λεπτομέρειες, αλλά η πρώτη μου αντίδραση είναι η εξής. Ορισμένοι από τους τομείς που εξετάζουμε στα πλαίσια ε, των, της μεγάλης εκμετάλλευσης δεν είναι καλά οργανωμένοι Η γεωργία, οι οικιακές εργασίες, συνεπώς η επίδραση ε, των μεταρρυθμίσεων της εργατικής νομοθεσίας σε αυτούς τους τομείς ε, θα είναι κάτι το πολύ δύσκολο και ο κύριος Λόπες αναφέρθηκε στα οικονομικά και κοινωνικά δικαιώματα συμφωνώ απόλυτα. Η χάρτα για τα θεμελιώδη δικαιώματα προβλέπει ίσους όρους σε όλα αυτά τα άτομα. Το κάθε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει υπογράψει ε, αυτό το σύμφωνο των Ηνωμένων Εθνών. Συνεπώς ο οργανισμός μας είναι υπεύθυνο απέναντι στα θεμελιώδη δικαιώματα και δεν μπορούμε να προχωρήσουμε αν δεν αναγνωρίσουμε ε, ίσα δικαιώματα, οικονομικά και θεμελιώδη σε όλους. Τέλος κύριε Μαρτά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Πράγματι είναι αδύνατον να γίνει σοβαρή ανάλυση καταστάσεων όπως αυτή χωρίς να λάβουμε υπόψη τα δύο φύλλα. Πάντοτε η θέση των γυναικών είναι διαφορετική και δυστυχώ μερικέ φορέ είναι χειρότερη από εκείνη των ανδρών. Αυτό πρέπει να το αναγνωρίσουμε στη μεθοδολογία που χρησιμοποιούμε. Επίσης συμφωνώ ε, για το ρόλο των συνδικάτων που είναι πολύ σημαντικός. Τα συνδικάτα παίζουν ζωτική σημασία ρόλο ε, για να υπάρχει μια υγιής κοινωνία των πολιτών στην Ευρώπη και θα πρέπει να υποφεληθούμε κάθε ευκαιρία να υποστηρίξουμε τα συνδικάτα. Και θα πρέπει λοιπόν ο ρόλος τους να είναι ελεύθερος. Μπορεί ο συνάδελφός μου να απαντήσει ορισμένα από τα ερωτήματα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να αναφερθώ σε κάποια από τα σημεία τα οποία θίξατε στις ερωτήσεις σας. Ο ρόλος της διευκόλυνσης, της επιχειρηματικότητας σε σχέση με το οργανωμένο έγκλημα. Δύο πράγματα θέλω να πω. Βεβαίως, η διακίνηση ανθρώπων, το λαθρεμπόριο, σίγουρα έχει εξεταστεί. Βλέπουμε όμως ότι αυτό δεν έχει γίνει και με κάποιες άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες και συμβατικές σχέσεις. Αυτό θα πρέπει να γίνει. Να γνωρίσουμε δηλαδή καλύτερα να υπάρξει έρευνα αυτών των τομέων και να δούμε πώς ακριβώς είναι οργανωμένες αυτές οι δραστηριότητες εκεί. Αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι δημιουργούμε την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος, όχι μόνο για τη διακίνηση, αλλά για κάθε είδος εκμετάλλευσης που μπορεί να συμβαίνει. Και θα πρέπει εδώ να προετοιμάσουμε τις εντολές όλων των ε, αστυνομικών δυνάμεων για να μπορέσουν να καταπολεμήσουν με αποτελεσματικό τρόπο κάθε είδους εκμετάλλευση και εγκληματική δραστηριότητα. Επαναλαμβάνω, δηλαδή και τη διακίνηση ανθρώπων και την εκμετάλλευση, την καταναγκαστική εργασία και όλες αυτές τις μορφές εκμετάλλευσης μέσω της εργασίας που φυσικά ε, γνωρίζουμε σήμερα ότι συμβαίνουν. Εκμετάλλευση μεταναστών. Τις περισσότερες φορές διαπιστώνουμε ότι επιχειρήσεις, γνωστές, ε, μεγάλοι όμιλοι χρησιμοποιούν μετανάστες, συμμετέχουν δηλαδή σε αυτήν την εκμετάλλευση. Και είναι νομική ευθύνη του εργοδότη, των επιχειρήσεων, εάν κάτι τέτοιο συμβαίνει. Κάθε φορά λοιπόν που εξετάζουμε την νομοθεσία των κρατών μελών διαπιστώνουμε ότι από νομικής απόψεως υπάρχουν τα εργαλεία για να παταχθεί αυτή η εκμετάλλευση. Πολλές φορές λοιπόν μιλάμε για πιθανές κυρώσεις, όπως παραδείγματο χάρη η δημοσίευση του καταλόγου των επιχειρήσεων αυτών που έχουν καταδικαστεί για εκμετάλλευση εργαζομένων κτλ. κτλ. Όλα αυτά λοιπόν τα εργαλεία τα οποία σε μεγάλο βαθμό τα διαθέτουμε θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για να παταχθούν αυτά τα φαινόμενα. Η υλοποίηση λοιπόν, η εφαρμογή αυτών που υπάρχουν είναι πιο σημαντικοί από το να ε, συζητάμε για τη δημιουργία νέων εργαλείων, νέων νομοθετικών ε, διατάξεων για την ε, πάταξη αυτών των φαινομένων. Ο πολύ σημαντικός ρόλος των συνδικαλιστικών οργανώσεων επίσης είναι κάτι που θίξατε στις ερωτήσεις σας οι βέλτιστες πρακτικές, η καθοδήγηση των εργαζομένων, η καλύτερη συνεργασία μεταξύ των ε, φορέων. Και βεβαίως το θέμα των ε, εξουσιών και αρμοδιοτήτων των συνδικαλιστικών οργανώσεων. Στη Δανία έχουμε πολύ συγκεκριμένο πλαίσιο που καθορίζει τις ε, αρμοδιότητες ε, και τις εξουσίες των συνδικαλιστικών οργανώσεων. Το θέμα της καθοδήγησης, το θέμα της ενημέρωσης προς τους εργαζόμενους. Είναι ένας καθοριστικός ρόλος που παίζουν ή θα έπρεπε να παίζουν ε, οι συνδικαλιστικές οργανώσεις. Ο ρόλος των γυναικών οι γυναίκες βεβαίως είναι θύματα και δεν είναι εύκολο πολλές φορές να αποδεχθούν ε, οι εργαζόμενοι ότι είναι θύματα. Και αυτό συμβαίνει βεβαίως κυρίως για τους άντρες εργαζόμενους. Ε, είναι πάρα πολύ σημαντικό για αυτούς η εικόνα τους, η εικόνα τους ε, για την οικογένειά τους που έχει παραμείνει στην ε, χώρα από την οποία προέρχονται. Είναι λοιπόν πολύ δύσκολο να αποδεχθούν ότι είναι θύματα εκμετάλλευσης. Ευχαριστώ πολύ. Οι περισσότερες ερωτήσεις έχουν απαντηθεί. Θα συμπληρώσω λοιπόν με κάποιες παρατηρήσεις. Προσπαθούμε να δημιουργήσουμε βάσει των εκτιμήσεών μας μία βάση εκκίνησης. Ποιες είναι οι γενικές τάσεις, παραδείγματος χάρη. Για να σας πω αν σήμερα, σε σχέση με την προηγούμενη δεκαετία, η εκμετάλλευση αφορά περισσότερους ή λιγότερους εργαζόμενους, θα πρέπει να έχω πολύ συγκεκριμένα στοιχεία, τα οποία σήμερα δεν διαθέτω. Ζητούμε λοιπόν τη συνεργασία των κρατών μελών για να μπορέσουμε να αποκτήσουμε συγκρίσιμα στοιχεία και το πρόβλημα είναι ότι συζητάμε για τη δημιουργία νέων νομοθετικών πλαισίων, νέας νομοθεσίας, ενώ σήμερα οι νόμοι και τα εργαλεία που διαθέτουμε δεν τα χρησιμοποιούμε, δεν τα ε, υλοποιούμε και δεν τα εφαρμόζουμε. Ένα θύμα βεβαίως μπορεί να προσφύγει στη δικαιοσύνη, ένα θύμα εκμετάλλευσης, για να ζητήσει να τηρούνται τα δικαιώματά του. Και βεβαίως είναι πάρα πολύ σημαντικό εδώ να υπάρχει συνεννόηση, ενημέρωση και να μεταφέρονται οι βέλτιστες πρακτικές από τη μία χώρα στην άλλη. Πρέπει επίσης ε, όλοι να εξετάσετε τις περιπτώσεις των ε, ε, εργαζόμενων οι οποίοι έπεσαν θύματα εκμετάλλευσης, τα οποία ε, υποθέσεις οι οποίες έχουν ε, σήμερα γίνει γνωστές, ε, οι εργαζόμενοι έχουν προσφύγει και υπήρξαν και αποζημιώσεις. Αυτές οι υποθέσεις πρέπει να γίνονται γνωστές, πρέπει να δημοσιεύονται. σα ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ ενδιαφέρουσα ήταν αυτή η συζήτηση. Βεβαίως είναι πάντα πολύ σημαντικό να υλοποιούμε και να εφαρμόζουμε τους υπάρχοντες νόμους, την υπάρχουσα νομοθεσία. Θα διακόψουμε για πέντε λεπτά πριν να περάσουμε στην ψηφοφορία στις 10. Υπότιτλοι So, colleagues, um, we can proceed with the votes now. Αρχίσουμε την ψηφοφορία. Cards, ready to go. Έχετε κάρτες ψηφοφορίας, μπορείτε να... Μπορούμε να ξεκινήσουμε. Πρώτη έκθεση, ρομποτική. ψηφίζουμε για τη συμβαστική 1. Τέσσερις, τέσσερις πολιτικέ πολιτικές, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 2. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Μετά, τροπολογία 14. Υπέρ, κατά, απορρίπτεται να έχουμε χωριστή ψηφοφορία στην τροπολογία 16. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά. Θα ζητήσω να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία για το πρώτο τμήμα της 16. Ψήφισατε όλοι. Περάς. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα της 16 υπέρ. Κατά αποχές. Νομίζω θα πρέπει να το λέξουμε και αυτό. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τώρα πάμε στη συμβαστική πρόταση 3. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 18 υπέρ κατά απορρίπτεται πάμε τώρα στη συμβαστική 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Σαράντα. τροπολογία 40 υπέρ κατά, αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 5 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 6 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 50 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 51 υπέρ. Κατά αποχές και αυτή εγκρίνεται. Συμβιβαστική 7 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 61 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Τώρα πάμε στη συμβαστική 8 υπέρ κατά άποχες εγκρίνεται 68 υπέρ κατά άποχες εγκρίνεται 71 υπέρ κατά άποχες απορρίπτεται 74 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται, 76 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται, 77 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Να ελέξουμε για την 77. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρα τη ψηφοφορία για την 77. Απορρίπτεται. «78. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική 9. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 10. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. 94. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. Έχουμε χωριστή ψηφοφορία στην 96 για το πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Θα λέω ότι και αυτή εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Θα ελέγξουμε. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά για το τρίτο τμήμα της 96. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 97 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 98 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά για την 98 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας για την 98 εγκρίνεται. 99 υπέρ κατά αποχές θα ελέγξουμε ψηφίζουμε ηλεκτρονικά για την 99 άρχεται Ψήφισατε όλοι. Πέρασε. Εγκρίνεται. Ψήφισμε τώρα τελική ψήφος. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Με μεγάλη πλειοψηφία εγκρίνεται. Now we move to the establishment of the structural reform support program. διαρθρωτικές ε, μεταρρυθμίσεις για το πρόγραμμα 17-20. Επόμενη ψηφοφορία. So the first vote is... Ψηφίζουμε πρώτα 58 και 59 τροπολογίες που είναι ταυτόσιμες, δηλαδή θέλουν να απορρίψουν όλη την ε, πρόταση. Ποιος είναι υπέρ, κατά, απορρίπτονται. Τώρα πάμε στην τροπολογία 187. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 188. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική U υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 191 τροπολογία υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 192 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 193 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 195 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται να ελέγξουμε ελέγχουμε ψηφίζουμε για το 195 πέρας της ψηφοφορίας απορρίφθηκε όντως 196 μία αποδεκτή πάμε στα 197 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 198 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 199 αποσύρθηκε 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 200 υπέρ κατά αποχές Απορρίπτεται. 20. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Θα ελέξουμε. Θα ελέξουμε. Νομίζω απορρίφθηκε, αλλά θα ελέξουμε, λέει Πρόεδρος. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβαστική Β. Υπέρ, κατά, άποχες, εγκρίνεται. Συμβαστική W. Υπέρ, κατά, άποχες, εγκρίνεται. 23. Υπέρ, κατά, άποχες, εγκρίνεται. 24 υπέρ κατά άποχες εγκρίνεται 203 υπέρ κατά άποχες θα ελέγξουμε 203 άρχεται πέρας γιατί 203 να εγκρίνεται με μεγάλη διαφορά 25 υπέρ κατά άποχες εγκρίνεται 204 υπέρ κατά άποχες ελέγχουμε για 204 ψηφίζουμε ηλεκτρονικά 204 204 ψηφίζουμε Πέρας. Απορρίπτεται. 205. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική X. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 211. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική Y, Y, υπέρ, κατά, εποχές, εγκρίνεται. 214. Υπάρχει προφορική τροπολογία για την 214, λέει ο Πρόεδρος. ναι, Πρόεδρε καταθέτουμε προφορική αντί για social well-being να πούμε social cohesion, κοινωνική συνοχή αντί για κοινωνική ευημερία. Υπάρχουν αντιρρήσει για αυτή την προφορική τροποποίηση. Όχι, ωραία, τη θέτουμε σε ψηφοφορία. Ποιος είναι υπέρ. Θα ζητήσω να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά, λέει ο πρόεδρο. Δεν ήταν ε, σαφέ το αποτέλεσμα. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Διακόσια Υπέρ. Κατά. Αποχές Νομίζω ότι απορρίφθηκε. Ωραία, να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά, λέει πρόεδρος. Άρχεται η ψηφοφορία για την 215 τροπολογία. Ψήφισατε όλοι. Πέρας. Απορρίφθηκε όντω. 216. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 217 υπέρ, κατά, άποχες, εγκρίνεται. 218 υπέρ, κατά, άποχες, απορρίπτεται. 219 καταπίπτει. 220 υπέρ, κατά, άποχες, απορρίπτεται. 221 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 222 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 223 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική ζήτα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική αλφα-αλφα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική ΑΙ υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική ΑΒ υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 234 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Να ελέγξουμε. Ωραία. για την 234 ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 235 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 30 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 236 καταπίπτει 237 και αυτή καταπίπτει όχι θα ψηφίσουμε λέει πρόεδρος για 237 υπέρ Κατά. Θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά για την 237. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. Περνάμε τώρα στην 238 με προφορική τροπολογία ως προσθήκη αντιρρήσει. Ωραία, θα ψηφίσουμε. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά για την 238. Ψηφίζουμε. Πέρα Απορρίπτεται. 239 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 240 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 241 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική AC υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 243 υπέρ. Κατά. Αποχές να απορρίπτεται. 32 και 244 μαζί. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 33 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 245 αποσύρθηκε, οπότε πάμε στη 34. 34 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 35 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 246 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 247 υπέρ. Κατά παχές, Εγκρίνεται. Συμβαστική AD. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική AH. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 254 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται, 255 υπέρ κατά αποχές θα ελέγξουμε ψηφίσουμε ηλεκτρονικά για 255 άρχεται η ψηφοφορία πέρας απορρίπτεται Amendment 256 in favor 256 υπέρ κατά αποχές Ελέγχουμε. Αρχή της ψηφοφορίας. Τέλος. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική ΑΕ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 2.59. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 2,60 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 2,61 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική αφ Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Α, συμβιβαστική υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 267 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 38 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 2,68 υπέρ, 2,68 υπέρ. Κατά. Αποχές. Να ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Δεν ξέρω γιατί. Αρχή της ψηφοφορίας. Τέλος. Απορρίπτεται. Εντάξει. 269, η 70 έχει αποσυρθεί. 269 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται νομίζω. 39 υπέρ. 39 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 271 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 2,72 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 2,73 υπέρ, κατά, αποχές. Νομίζω ότι πρέπει να ελέγξουμε τη 2,73 αρχή της ψηφοφορίας. Τέλος. Απορρίπτεται. 2,74 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται, 2,75 υπέρ, κατά, αποχές, ελέγχουμε ηλεκτρονικά, 2,75, αρχή της ψηφοφορίας. Τέλος. Απορρίπτεται. 40. Τροπολογία 40 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 2.76 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 2.77 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Περνάμε στην τροπολογία 41 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 2,79 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 42 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 43 υπέρ κατά αποχές ελέγχουμε. Την 43. Ψηφίζουμε. Ένας παραπάνω ψηφίζει από το ΕΛΚ. Όχι. Τώρα είμαστε εντάξει. Εγκρίνεται. Τροπολογία 281 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ελέγχουμε. Αρχή της ψηφοφορίας 281. Τέλος. Απορρίπτεται με μεγάλη πλειοψηφία. AJ, συμβιβαστική, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 283 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 284 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 285 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 286 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 287 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 44 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική AG υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 46 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 289. Όχι. Δεν ψηφίζουμε τη 289. Η επόμενη τροπολογία που ψηφίζουμε είναι 2.92. Όχι. Η τροπολογία 50. Λέει η πρόεδρος. Είναι η επόμενη. Δεν ψηφίζουμε τη 289, γιατί εγκρίθηκε η 287. Δεν εγκρίθηκε η 287, άρα Η επόμενη τροπολογία που θα ψηφίσουμε είναι η 50. Συμφωνείτε υπέρ. 50. Τροπολογία 50 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 51. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 294 έχει αποσυρθεί, 295 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Κατόπιν ψηφίζουμε συνολικά την 52, 53, 54 και 56 υπέρ. Κατά αποχές θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Αρχή της ψηφοφορίας. Τέλος, εγκρίνονται. 2,96 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνονται. 2,98 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 2,99 Η 53 έχει ψηφιστεί. Ψηφίζουμε την τροπολογία 299 υπέρ. Ναι. Άρα πρόκειται για την 299. Αποχές. Εγκρίνεται η 299. Και τώρα ψηφίζουμε την τροπολογία 57. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Αιτιολογικές σκέψει. Συμβιβαστική G. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Αιτιολογική 63 δεν είναι αποδεκτή. Τροπολογία 64 με την προφορική υποτροπολογία υπέρ κατά αποχές ελέγχουμε την τροπολογία 64 αρχή της ψηφοφορίας τέλος απορρίπτεται 65 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 2 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική α υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 73 και 74 από κοινού υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτονται. Συμβιβαστική Β υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 8 δεν είναι αποδεκτή. 81 υπέρ κατά αποχές Νομίζω ότι πέρασε. Συμβιβαστική ε, υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 83 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική C υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 91 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική D υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 101 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική F υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Περνάμε στην τροπολογία 109 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 110 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβιβαστική H υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική I, Ι, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. περνάμε στην τροπολογία 126. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική J. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική N, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική R, ρο, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 135 υπέρ. Κατά. Αποχές. Α, δεν ψηφίζουμε. Δεν ψηφίζουμε την 135. 136 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβεβαστική κάπα. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. περνάμε στην τροπολογία 142 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 143 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική L λάμδα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Περνάμε στην 146 υπέρ κατά αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική αίμα, μη, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. «156 και 157 από κοινού υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτονται. Συμβαστική ο, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 161 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική π υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 166 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική Q υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 169 υπέρ κατά αποχές, απορρίπτεται. 170 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 171 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 177 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβιβαστική Σ, σίγμα, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 180 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 183 υπέρ. Α, όχι, συγγνώμη, λέει ο Πρόεδρος. 182 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 183 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική ταφ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 185 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Και τώρα ψηφίζουμε την τελική ψηφοφορία του κειμένου. Αρχή της ψηφοφορίας. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος. Εγκρίνεται Και τώρα περνάμε στην ψηφοφορία για το Εράσμος Plus. Συμβαστική Α υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική Β υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική ο, όμικρο, υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 25, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται, 25. Συμβιβαστική ταφ, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική S, σίγμα, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική Q υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 32 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική N, νη, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική B, υπέρ. Α, υποτροπολογία προφορική. Είναι κάποιος κατά, όχι. Ψηφίζουμε τη Β λοιπόν. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική Σ υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική ρο υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική G υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Θέλετε να ελέγξουμε? Αρχή της ψηφοφορίας συμβιβαστική G. Τέλος. Εγκρίνεται με μεγάλη πλειοψηφία. Συμβιβαστική έλα, λάμδα, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 53 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 54 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική γιώτα, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 56. Δύο τμήματα. Το πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, ελέγχουμε ηλεκτρονικά το δεύτερο τμήμα της 56. Τέλος, απορρίπτεται. Περνάμε στην συμβαστική F υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 62 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίζουμε την 62. Τέλος. Απορρίπτεται η 62. 63 υπέρ κατά αποχές απορρίψετε. Συμβαστική D υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 78 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική K υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική ε υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική π υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 95 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 98 υπέρ, κατά, αποχές, Ελέγχουμε ηλεκτρονικά την 98. Τέλος. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική H. Υπέρ, κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 103 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 104 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 105 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 108 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 114 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 115 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 1. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 118 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 125 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 127 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική γιου, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 137 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 138 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 139 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 140 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 146 υπέρ, κατά, αποχές ψηφίζουμε ηλεκτρονικά την 146 αρχή της ψηφοφορίας. Τέλος. Εγκρίνεται. 148 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Περνάμε στις τελειολογικές σκέψεις. Τροπολογία 1. Υπέρ. Α, να τις ψηφίσουμε όλες μαζί. Από τη 1 έως τις, την 7 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνονται. Οκτώ υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Εννιά κατά, αποχές, εγκρίνεται. Και τώρα κάνουμε την τελική ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Αρχή της ψηφοφορίας. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος. Και βεβαίως εγκρίνεται με πολύ μεγάλη πλειοψηφία. Now we move to the question for all. Περνάμε στην ερώτηση, η προφορική απάντηση, το θέμα της εγγύησης των, ε, αρμοδιοτήτων, των δεξιοτήτων, συγγνώμη, συμβαστικό κείμενο υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται και τώρα όλα τα άλλα καταπίπτουν και πάμε στην τελική ηλεκτρονική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε. Μεγάλη πλειοψηφία, εγκρίθηκε το κείμενο και θα περάσει από την Ολομέλεια του Νοεμβρίου.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 Uh, λοιπόν, το επόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη είναι από την uh, Επιτροπή σε σχέση με την κατεξοδότηση πράξη και κατόπιν έχουμε τη συνέχεια uh, στην Ευρωπαϊκή Εκδήλωση Νεολαίας. Σε αυτή την αίθουσα λοιπόν υπάρχουν περίπου 210 θέσεις και υπάρχουν 100 νέοι περίπου που θα έρθουν κοντά μας. Θα ήθελα να παρακαλέσω τα μέλη λοιπόν και το προσωπικό να προχωρήσουν στα μπροστινά καθίσματα και όποια μέλη θα έρθουν ε, θα είναι καλοδεχούμενοι, αλλά κόλλα θα ήταν να κάνουμε χώρο στους νέους, προκειμένου τα 100 άτομα που θα έρθουν, οι νέοι που θα έρθουν, να έχουν άδεια καθίσματα, να μπορούν να βρεθούν κοντά μα. Γι' αυτό παρακαλώ να προχωρήσετε στα μπροστινά καθίσματα, αν γίνεται, για να τους αφήσουμε τι πίσω θέσει άδειε. Βεβαίω. Ε, είναι δύσκολο αν έχουν ονόματα μπροστά σα Γι' αυτό θα σας παρακαλούσα να συμπληρώσετε τα κενά καθίσματα και να αφήσετε όσο γίνεται κενά καθίσματα στις πίσω σειρές. Okay, so our next item... Το επόμενο θέμα λοιπόν είναι πολύ τεχνικό τεχνικό από την Επιτροπή και είναι ο κατουξιδός το κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και αφορά την απλούστευση για τον υπολογισμό ε, των επιστροφών που γίνονται, επιστροφών δαπανών των κρατών μελών. Παρακαλώ την κυρία Αντριάννα Σουπόβα να μας παρουσιάσει το θέμα. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Το άρθρο 41 του κανονισμού επιτρέπει στην Επιτροπή να υιοθετήσει κατεξοδόση κανονισμό ε, για το μοναδίο κόστης που αποτελεί βάση για την επιστροφή των δαπανών των κρατών μελών από την Επιτροπή. Και επιτρέπει επίσης να προσαρμόζονται αυτά τα αιτήματα χωρίς να συζητηθεί περαιτέρω με την Επιτροπή. Αυτή είναι η πρώτη φορά που παρουσιάζουμε παραρτήματα σε αυτό το κατσουδότσι κανονισμό και ο στόχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφέρθηκε πρόσφατα. Θέλουμε να εστιάσουμε όλες μας τις προσπάθειες στην επίτευξη αποτελεσμάτων με βάση απλουστευμένες διαδικασίες και απλουστευμένες δαπάνες για την επιστροφή, προκειμένου τα κράτη-μέλη να εστιάζουν τις προσπάθειές τους για την επίτευξη των καλύτερων αποτελεσμάτων στα πλαίσια των χρημάτων που υπάρχουν στον προπολογισμό. Υπάρχουν πολλά θετικά σημεία όσον αφορά αυτό το απλουστευμένο σύστημα για ορισμένα κράτη-μέλη και για ορισμένες ε, λειτουργίες. Και αυτό δίνει μια νομική ασφάλεια στα κράτη-μέλη, ώστε να μην υπάρχουν ε, δυσκολίες, διότι πρέπει να προσπαθούμε να ακολουθούμε μια μεθοδολογία, ε, περιορίζουμε ε, τη δουλειά των ελεγκτών και έχουμε ένα σωστό προσανατολισμό και επίσης μπορούμε να εφαρμόσουμε αυτές τις δαπάνες σε λειτουργίες που έχουν σχέση με διαγωνισμούς, δημόσιους διαγωνισμούς. Τα βασικά στοιχεία αυτής της απλουστευμένης διαδικασίας υιοθετεί τυποποιημένους κανονισμούς σύμφωνα με το άρθρο 41 και αποτελεί τη βάση για την επιστροφή στα κράτη-μέλη των δαπανών που έχουν σχέση με την εφαρμογή των επιχειρησιακών προγραμμάτων. όσον αφορά τις σχέσεις μεταξύ ε, των διαχειριστικών αρχών ε, και των αποδεκτών. Γι' αυτό πρέπει να δούμε πώς γίνεται η πιστοποίηση των δαπανών και οι διαχειριστικές αρχές στέλνουν τις απαιτήσει με βάση την απλουστευμένη διαδικασία όσον αφορά τις δαπάνες που έχουν συμφωνηθεί στα πλαίσια του κανονισμού. Τα κράτη-μέλη μπορούν να εφαρμόσουν τις δικές τους λογιστικές μεθόδους και συμφωνήσαμε ότι όταν το ζητήσει ένα κράτος μέλος να προσαρμόσουμε κάθε χρόνο αυτές ε, ε τις απλουστευμένες ε, διαδικασίες χωρίς να χρειάζονται προηγούμενα δικαιολογητικά. Το μόνο αρνητικό στοιχείο είναι ότι προς το παρόν αυτή η απλούστευση αφορά τις διαδικασίες του ESF και όχι τις άλλες. Όπως είπα πρωτήτερα, αυτός ο κατουξιδός κανονισμός υιοθετήθηκε τον Ιούλιο του 2015 και το βασικά καλύπτει τις διαδικασίες των λειτουργιών, τον ορισμό και τα ποσά καθώς και τις προσαρμογές. Τα παραρτήματα προσαρτώνται κάθε φορά που υπάρχουν επιπλέον αιτήματα από τα κράτη-μέλη για να συζητήσουμε ορισμένα επίπεδα μονα, ε, μοναδίων δαπανών και προσαρτώνται αυτά τα παραρτήματα ε, στον κατεξουδότηση κανονισμό. Επειδή ο κατεξουδότηση κανονισμός καλύπτει μόνο τη Γαλλία και τη Σουηδία, επειδή είναι τα μόνα κράτη-μέλη τα οποία εφαρμόζουν τις τα δαπάνες, Για τη Γαλλία είχαμε συμφωνήσει να καλύψουμε δαπάνε και για τη Σουηδία ορισμένε δαπάνε και αμοιβέ συμμετεχόντων που καλύφθηκαν σε ορισμένου τομεί προτεραιότητα. Η πρώτη τροπολογία αυτού του κανονισμού υιοθετήθηκε στις 18 Μαρτίου 2016. Γι' αυτό δεν αλλάζουμε τα άρθρα του αρχικού κανονισμού, αλλά ε, προσθέτουμε δύο νέα παραρτήματα για το Βέλγιο και την Τσεχική Δημοκρατία, για την οποία έχουμε πέντε μοναδιές δαπάνες που καλύπτουν την αύξηση των προμηθειών για τις εγκαταστάσεις φροντίδας του παιδιού και το Βέλγιο δύο μονάδες. η νέα τροπολογία που παρουσιάζω στο άρθρο 14.1 καλύπτει επιπλέον μοναδιές δαπάνες για την Τσεχία και νέες μοναδιές δαπάνες για τα κράτη-μέλη που είναι η Σλοβακία, η Μάλτα, η Ολλανδία και η Ιταλία και η Δανία. Για την Τσεχική Δημοκρατία έχουμε δύο τομείς όπου έχουν συμφωνηθεί αυτές οι απλουστευμένες δαπάνες και επίσης υποστήριξε φοιτητές ε, και ε, στο προσωπικό εκπαιδευτικών εγκαταστάσεων. Εδώ έχουμε 12 μονάδες. Επίσης το παράρτημα αφορά και την φροντίδα του παιδιού που είχε ήδη υιοθετηθεί στην προηγούμενη τροπολογία στον κανονισμό σύμφωνα με το επιχειρησιακό πρόγραμμα και θα εφαρμοστεί για το, πρόγραμμα, το επιχειρησιακό πρόγραμμα για την Πράγα. Επίσης, Έχουμε μοναδιές δαπάνες για την κατάρτιση των υπαλλήλων με βάση το κόστος και την έρευνα της αγοράς. Τώρα, όσον αφορά την υποστήριξη στην εκπαίδευση, χρησιμοποιούμε επίσημες στατιστικές μισθολογίων για τον τομέα της εκπαίδευσης και αυτές οι μοναδιαίες τιμές θα καλύψουν 400 εκατομμύρια ευρώ στα πλαίσια των επιχειρησιακών προγραμμάτων. Πάντοτε για την τσεχική δημοκρατία. Για τη Μάλτα, το επόμενο παράρτημα, συμφωνήσαμε να βοηθήσουμε τους μειονεκτούντες εργαζόμενους και εκείνους που έχουν αναπηρία με βάση τα ποσοστά του χαμηλότερου συντελεστή ε, του Εθνικού Μισθολογίου. Και αυτό θα καλύψει περίπου 10 εκατομμύρια ευρώ σε δαπάνες πάλι μπορούν να προσαρμοστούν ανάλογα με τις αλλαγές σύμφωνα με τους ελάχιστους μισθούς στη χώρα. Για την Ιταλία τώρα. Έχουμε ένα μεγάλο παράρτημα για αυτή τη χώρα επειδή καλύπτει δύο βασικές περιοχές. Πρώτα απ' όλα το επιχειριακό πρόγραμμα Εθνικής Εμβέλειας και την υποστήριξη για υποτροφίες, για έρευνα που καλύπτονται από εθνικά και, και περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα χρησιμοποίησαμε περιφερειακά δεδομένα για παρόμοιες ε, επιχειρήσεις σε προηγούμενες περιόδους, καθώς και ενωσιακά ποσοστά κινητικότητας για, ε, για το επίπεδο PhD ε, οι δαπάνες βασίζονταν στο, στα εθνικά τιμολόγια. Η προσαρμογή τώρα για την Ιταλία όσον αφορά το δίκτυο του καταναλωτή είναι τη τάξη του 5%. Εάν υπάρχουν αλλαγές ανάλογα με του εθνικού ε, ε, κανονισμού, πάλι χρειάζεται ε, μια προσαρμογή. Προβλέπεται ότι αυτή η προσαρμογή διαδικασία θα καλύψει 900 εκατομμύρια ευρώ στην Ιταλία. Για τη Σλοβακία τώρα, Έχουμε δύο δαπάνες για τις ξένες γλώσσες και για τις δεξιότητες σε επικοινωνία και πληροφορική. Επίσης για παιδικούς σταθμούς και ε, δημοτικά και το, τα μοναδιές δαπάνες καλύπτουν άμεσες δαπάνες ε, για εκπαίδευση θα υπάρχουν περίπου 80 εκατομμύρια ευρώ που θα δαπανηθούν με την χρησιμοποίηση αυτής της απλουστευμένης διαδικασίας. Για τη Γερμανία τώρα, που είναι η πρώτη περιοχή του Mecklenburg-Verbommen, όπου έγινε η πρόταση για εννέα κόστη που συνδέονται με την ανάπτυξη αυτών των ενταξιακών σχολείων. Ο στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα σύστημα ενταξιακών σχολείων και να μειωθεί η ανάγκη για ειδικά σχολεία. Όλα αυτά αφορά την ε, εκπαίδευση των δασκάλων και επίσης ε, αυτό θα καλύψει 14 εκατομμύρια ευρώ που θα δαπανηθούν στα πλαίσια της χρησιμοποίησης αυτής της διαδικασίας και δεν έγινε έτοιμα για προσαρμογή της μεθόδου. Εάν η περιοχή εκείνη της Γερμανίας αποφασίσει ότι αυτές οι, οι μοναδίες δεν είναι ρεαλιστικές, μπορούν να αναδιαπραγματευτούν το επίπεδο των δαπανών. Τελευταίο κράτος μέλος που ζήτησε τις μοναδίε δαπάνε είναι η Ολλανδία. Υπάρχουν τρεις μοναδίε δαπάνε όσον αφορά δραστηριότητε επανένταξη για τους κρατούμενους ε, και για νέου που βρίσκονται σε ιδρύματα. Η πληρωμή θα βασιστεί στον αριθμό των ημερών παρέμβαση. Τα ποσά θα βασίζονται στι συνολικέ δαπάνε των υπηρεσιών και των προηγούμενων προγραμμάτων και στον συνολικό αριθμό των ημερών παρέμβαση. Και τα ποσά θα προσαρμοστούν ετησίως σύμφωνα με τον δίκτυ καταναλωτή της χώρας και θα καλύψουν περίπου 43 εκατομμύρια ευρώ. Ως συμπέρασμα, θέλω να σας πω ότι υπάρχει όλο και των ενδιαφέρων... για αυτή τη δυνατότητα εφαρμογής του άρθρου 14 παράγραφος 1. Μέχρι τώρα αυτή η διαδικασία υιοθετήθηκε ως παραρτήματα στον κατασκευαστικό κανονισμό και καλύπτει 2,9 δις ευρώ και συνεργαζόμαστε με τα κράτη-μέλη και υπάρχουν ενεξελίξει νέες προτάσεις για να δούμε άλλες δυνατότητες εφαρμογής αυτής μεθόδου. Επίσης έχει δεσμευθεί Επιτροπή να εφαρμόσει σε νοσιακό επίπεδο αυτή τη μέθοδο που θα εφαρμόζεται σε όλα τα κράτη-μέλη αλλά δεν χρειάζεται να δικαιολογηθούν, δεν θα εξετάσουμε άλλες μεθοδολογίες, αλλά θα συνεχιστεί η εργασία που γίνεται από την ομάδα υψηλού επίπεδου. Γι' αυτό η Επιτροπή θα προτείνει ενωσιακή μέθοδο. Συνεχίζονται οι προσπάθειές μας και ελπίζουμε ότι θα έχουμε έναν άλλο κατεξιδότη κανονισμό ενωσιακού επίπεδου και ότι τα κράτη-μέλη θα κάνουν προτάσεις που θα περιληφθούν ε, στον κατεξοδότηση κανονισμό του 2017. Ευχαριστώ πολύ. Thank you. Now Ευχαριστώ. Τα μέλη τώρα. Ο κύριος Λόπες, πρώτα. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Ερώτηση. Απλή. Πώς πιστεύετε ότι θα επηρεάσει την εφαρμογή αυτής της διαδικασίας της απλούστευσης το θέμα των εγγυήσεων για τους νέους, μιας και μιλάμε για ανεργία των νέων, που αφορά ιδιαίτερα χώρες όπως η Ισπανία, όπου έχουμε θέματα αφορολογικά, δημοσιονομικά, πειθαρχία κτλ. Αυτό πώς θα επηρεάσει το θέμα αυτού των νέων. Ευχαριστώ. Υποθέτω θα δούμε μία μείωση όσον αφορά τα λάθη που υποβάλλουν στα στοιχεία οι χώρες μέλη. Αυτό είναι καλό. Απλούστευση σημαίνει επίσης ότι μπορεί να έχουμε και αυστηρότερες προδιαγραφές υποβολής στοιχείων ώστε η απλούστευση να αφορά και άλλα στοιχεία. Αλλά θα ήθελα να μάθω κατά πόσο αυτή η απλούστευση θα περάσει και στους αποδέκτες του προγράμματος, ώστε να είναι οριζόντια, ώστε και αυτοί να υποβάλουν τους λογαριασμούς τους σωστά. Έχουμε λοιπόν κάτι το συλλογικό, ομαδικό και όχι κάτι το μεμονωμένο. Ισχύει και για αυτούς λοιπόν. Ευχαριστώ κύριο Σπρέντσικη. Ευχαριστώ πρόεδρε, ευχαριστώ. Ευχαριστώ την Κομισιόν για την πρόταση και για την ταχεία αντίδραση, για την απλούστευση. Εμείς πάντως θα θέλαμε να μειώσουμε και τις παρατυπίες και επιβεβαιώνω ότι στην Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού είχαμε μια ισχυρή σύσταση προς την Κομισιόν ώστε να προχωρήσει σε αυτή την κατεύθυνση. Όπως είπε η εκπρόσωπος της Κομισιόν σήμερα, βλέπουμε ότι υπάρχει μια συμβολή ήδη από τώρα. Ευχαριστώ. Χόκινγκ, επόμενη ομιλήτρια. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, ευχαριστώ την Επιτροπή. Συμφωνώ με τον προλαγήσαντα. Ευχαριστούμε την Κομισιόν που τελικά επέβαλε αυτή την πρόταση. Να ρωτήσω και να πω ότι είδαμε και την έκθεση του ελεκτικού συνεδρίου. Να ρωτήσω λοιπόν ποια είναι η δικιά τους η άποψη, τι κατευθυντήρες γραμμές έχουν προτείνει. Και όπως είπε και η Τζιν Λάμπερτ, αυτή η απλούστευση του κόστους. Συνεχώς ακούμε ως βουλευτές απόψεις σχέση με πρόσβαση σε κονδύλια της Ένωσης, γραφειοκρατία κτλ. Εγώ προσπαθώ να τα εξηγώ όλα αυτά και κάθε χρόνο εγκρίνουμε και ψηφίζουμε τον περιπολογισμό. Όλα αυτά πρέπει να είναι και αντισταθμιστικά. Γι' αυτό ακριβώς να ρωτήσω κι εγώ το ίδιο ερώτημα με την Τζιν. Αυτά επεκτείνονται, είναι οριζόντια. Δηλαδή μπορούμε να πούμε ότι εμείς ήδη κάνουμε κάτι το οποίο θα έχει σημασία για όλους τελικά και θα μας βοηθήσει στο να μειώσουμε τα λάθη όσον αφορά την υποβολή στοιχείων. Ευχαριστώ. Ο Τόμας Μάν, τελευταίος ομιλητής. Ευχαριστώ. Εγώ δεν ήθελα να πάρω το λόγο, αλλά τελικά είναι χρήσιμο να ακούει κανείς ε, τελικά ότι οι εκπρόσωποι τελείως διαφορετικών πολιτικών ομάδων έχουν τελικά τις ίδιες προτάσεις ή παρόμοιες προτάσεις. Το θέμα λοιπόν εδώ είναι αν πραγματικά οι λύσεις που προτείνονται ανταποκρίνονται στις προκλήσεις. Η απλοποίηση είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Και κάθε φορά βλέπουμε ότι οι προσπάθειες στον τομέα αυτό μας οδήγησαν σε απογοήτευση. Ελπίζω Ελπίζω κάτι να βγει από αυτήν την πρόταση και αν κάτι συγκεκριμένο από το οποίο μπορούμε να ξεκινήσουμε μπορεί να θεωρηθεί σαν εγγυημένο, τότε να βασιστούμε σε αυτό και να προχωρήσουμε. Βεβαίως και εδώ υπάρχει μια προστιθέμενη αξία από το ευρωπαϊκό επίπεδο. Και σίγουρα τα κέρδη από αυτό, τα ωφέλη από αυτό θα πρέπει να είναι απτά. Θα πρέπει να μπορούμε να τα δούμε και να τα αντιμετωπίσουμε σαν ε, ωφέλη για όλους μας. Thank you. Um, ευχαριστώ. Ακούσατε ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις που μοιάζουν. Κομισιόν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την υποστήριξη της δουλειάς μας για αυτή την απλουστευμένη διαδικασία επιλογών κόστους. Πράγματι, οι περισσότερες ε, χώρες που ανέπτυξαν αυτή τη διαδικασία την μεταβίβασαν στους τελικούς αποδόχους. Όχι μόνο δηλαδή σε σχέση με την Κομισιόν για την πιστοποίηση των δαπάνων κτλ. Για, τις μοναδιές, για το μοναδίο κόστος, αλλά και για τη χρήση των ίδιων μονάδων κόστους. Αυτό θεωρούμε ένα σημαντικό βήμα. Βέβαια δεν έχει γίνει πλήρως 100%. Να πω ότι πάντως οι χώρες αποφάσισαν ότι θέλουν την ίδια προσέγγιση, αλλά πολλές από τις μονάδες κόστους που υλοποιήθηκαν μέσω κανονισμού, πολλές από αυτές έχουν μετατοπιστεί, έχουν πάει και στους τελικούς αποδέκτες. Αξιολογούμε επίσης θετικά την ανακοίνωση του ελεκτικού συνεδρίου για την απροστευμένη χρήση αυτών των διαδικασιών, όπου δεν βλέπουμε παρατυπίες, δεν βλέπουμε διορθώσεις οικονομικές και αυτό προσφέρει κάποια σταθερότητα και για τις χώρες μέλη, όταν γνωρίζουν δηλαδή το ύψος του προπολογισμού και το πώς μπορούν να το χρησιμοποιήσουν. Τώρα, για τις εγγυήσεις και τις πρωτοβουλίες απασχόλησης στην Ισπανία, Χρησιμοποιήσαμε αυτές τις διαδικασίες, αλλά βέβαια λόγω περιπλοκότητας και διαφοράς μεταξύ περιφερειών είχαμε κάποιες προκλήσεις, πάντως δεν υποχωρήσαμε. Προσπαθούμε να αναπτύξουμε απλουστευμένες διαδικασίες κόστους που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν στην Ισπανία. Νομίζω ότι κάποια από τα εκπαιδευτικά μέτρα ιδιαίτερα που είναι πρώτης προτεραιότητας για μας για πανευρωπαϊκή δικασία, δηλαδή η απλούστευση κόστου, θα είναι διαθέσιμα και για την Ισπανία και θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν εύκολα από τη χώρα και σε όλες τις περιφέρειές της. Να χρησιμοποιηθούν δηλαδή όταν έχουμε λειτουργικά προγράμματα, συγγνώμη, επιχειρησιακά προγράμματα για την νεολαία. Οι ίδιες οι περιφέρειες της Ισπανίας κάνουν λιγότερους υπολογισμούς και ελέγχους για το κόστος. Αλλά βλέπουμε τελικά ότι από τη στιγμή που υπάρχει κατάρτιση για κάποιο άτομο υπάρχει άμεσα η καταβολή των κονδυλίων. Προς το παρόν λοιπόν δεν μπορούμε να πούμε ότι έχουμε σοβαρές επιπτώσεις όσον αφορά εφαρμογή των εγγύσεων για την Ισπανία γιατί αυτές οι επιλογές πιστοποιούνται βάσει του πραγματικού κόστους. Ευχαριστώ. Um, Ευχαριστώ πολύ. 15 πέμπτη Νοεμβρίου είναι η προθεσμία για υποβολή αντιρρήσεων και 31 Δεκεμβρίου στο Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ πολύ. Επόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη. Θα περιμένουμε στις 11.30 όμως για να ξεκινήσει είναι ακριβώς αυτή η συνοδευτική ακρόαση για την Ευρωπαϊκή Εκδόση για την Νεολαία. Μέχρι τι 11.30 λοιπόν θα περιμένουμε διάλειμμα.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 να καλύψουμε όλες τις κενές θέσεις. Jean, if you can come forward, that's great. Jean, έλα να καθίσει εδώ μπροστά. Φέρτε και το καρτελάκι σας μπροστά, να αφήσουμε τους χώρους στους νέους. Αν δεν έχετε καθίσει ακόμα, μπορείτε να βρείτε θέση εδώ μπροστά. Έχουμε αρκετές ε, κενές θέσεις. Um, Συνάδελφοι, ας ξεκινήσουμε. Θα έρθουν κι άλλοι, αλλά επειδή ήδη έχει περάσει η ώρα, για να μην χάνουμε χρόνο, να καλωσορίσω όλους τους επισκέπτες μας σήμερα. Έχουμε γύρω στους 100 νέους σήμερα. Ρίγα, Στρασβούργο, Λιέγη, από εκεί προέρχονται. Καλωσορίσατε όλοι σας και όλες σας. Now the, the second edition. Έχουμε τη δεύτερη έκδοση του EYIE e, που έγινε στο Στρασβούργο το Μάη φέτος με πάνω από 7.500 νέους που συζήτησαν ιδέες και προτάσεις για την αυριανή Ευρώπη. Η σημερινή λοιπόν ακρόαση αποτελεί ένα follow-up αυτής της εκδήλωσης του Στρασβούργου. Ταχεία εκδήλωση. Οπότε θα έχετε πολύ χρόνο και θα σας ζητήσω από τώρα να τηρήσετε το χρόνο ομιλία σας, αλλά με ιδιαίτερη χαρά καλωσορίζω τρεις συμμετέχοντες που ήρθαν σήμερα στην ακρόαση για να προσφυάσουν απόψεις για διάφορα ζητήματα όπως μετανάστευση και αγορά εργασίας, ανάπτυξη δεξιοτήτων ως μέσο αντιμετώπισης της ανεργίας των νέων και μετά νέοι επιχειρηματίες και startups. Θα κάνουμε λοιπόν ένα ideas check. Ένα σχήμα δηλαδή που αναπτύχθηκε για αυτού του είδους ακροάσεις. Θα ακούσουμε λοιπόν κάποιες ιδέες τρία προεπιλεγμένα μέλη θα απαντήσουν σε αυτές τις ιδέες. Έτσι το έχουμε σχεδιάσει. Να παρουσιάσω λοιπόν τους ομιλητές καταρχάς. Λόρας Νόινα από τη Γερμανία που θα μας παρουσιάσει ιδέες για την ανάπτυξη δεξιοτήτων ως μέσο αντιμετώπισης της ανεργίας των νέων και για τους νέους επιχειρηματίες και τις startups. Μελίσσα Τσίφκη από το Ηνωμένο Βασίλειο που θα μας παρουσιάσει ιδέες για τους μετανάστες και την αγορά εργασία και για τους νέους επιχειρηματίες και τις startups και μετά Λεόνι Σούλτς από τις κάτω χώρες που θα μας παρουσιάσει ιδέες για τους μετανάστες και την αγορά εργασία και την ανάπτυξη δεξιοτήτων ως τρόπος αντιμετώπισης ανεργίας πάντα. Έχουμε και ένα hashtag στο Twitter για αυτή την εκδήλωση, εκδήλωση EYE 2016 e με το hashtag μπροστά. Ελπίζαμε να έχουμε και λογαριασμό στο Twitter, αλλά δεν κατέστη δυνατό. Τέλο πάντων, δεν πειράζει. Μπορείτε να μπείτε όλοι στο Twitter και να μας παρακολουθήσετε από εκεί. Δύο λεπτά λοιπόν για κάθε ομιλητή EYE, e, δύο λεπτά για κάθε ευρωβουλευτή και μετά ένα λεπτό για δευτερολογία. Και στο τέλος, στο τέλος, θα έχουμε τον κύριο Σέρβο στο Γενικό Διευθυντή, ο οποίο θα απαντήσει εκ μέρους της Κομισιόν για αυτά που θα υποθούν. Είναι λοιπόν σημαντικό, ξαναλέω, να τηρήσουμε το χρόνο ομιλίας. Δεν θα πολύ χρησιμοποιήσω το σφυράκι, αλλά υπενθυμίζω και πάλι να τηρήσετε τους χρόνους. Πρώτος γύρος λοιπόν, για το θέμα των μεταναστών και της αγοράς εργασίας. Λέωνι Σούλτς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να επιταχύνει το θέμα της αναγνώρισης των διπλωμάτων, το θέμα της μετανάστευσης, για τους οποίους είναι απαραίτητο να δίνονται ευκαιρίες για την ενσωμάτωση στην αγορά απασχόλησης έτσι ώστε να μπορέσουν να ενσωματωθούν στις κοινωνίε μας. Χρειάζονται λοιπόν ευρωπαϊκά πρότυπα και η αναγνώριση των διπλωμάτων θα πρέπει να γίνεται με τον εξή τρόπο. Να μην υποχρεούνται να αποδείξουν τα διπλώματά τους στις ε, δεξιότητές τους και θα πρέπει να υπάρχει ένας ε, φορέας ο οποίος θα αναγνωρίζει τα διπλώματα καθώς και την εμπειρία την επαγγελματική τους αλλά και τις επαγγελματικές τους δεξιότητες. Αυτό θα πρέπει να γίνεται με έναν αντικειμενικό τρόπο και να παραμένει η προσεξέταση κατηγορία των ετούντων άσυλο χωρίς επαγγελματικές δεξιότητες. Επίσης συμπεριλαμβάνουμε και δύο παραγράφους για την διαφάνεια που θα πρέπει να επικρατεί όσον αφορά την αναγνώριση των διπλωμάτων για άτομα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στα πλαίσια της προσπάθειας ε, να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις ε, της παγκοσμιοποίησης, η Ευρωπαϊκή Ένωση καλείται να περιορίσει τον κοινωνικό αποκλεισμό, να ενσωματώσει τους ε, μετανάστες που φτάνουν σε εμάς με συγκεκριμένε επαγγελματικές δεξιότητες και να τους δώσει πρόσβαση στην αγορά εργασίας. Είναι κάτι καθοριστικό για τους μετανάστες έτσι ώστε να μπορέσουν να ενσωματωθούν και να γίνουν οικονομικά ανεξάρτητοι. Για τους πρόσφυγες ε, επίσης θα πρέπει να δίνεται η ευκαιρία να ενσωματώνονται στην οικονομία μας και στην κοινωνία μας. Οι άνθρωποι αυτοί είχαν μια ζωή πριν φτάσουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα πρέπει αυτή η ζωή και αυτή η εμπειρία να λαμβάνεται υπόψη και να μην τους υποχρεώνουμε να ξεκινήσουν από το μηδέν τη νέα του ζωή. Ευχαριστώ. Πάρα πολύ. Τώρα θα δώσω το λόγο σε εσά για δύο λεπτά επέκταση του νόμου για τις ευκαιρίες να υπάρχει μια ευρεία βάση δεδομένων που να λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες ε, των προσφύγων από κάθε χώρα. Βλέπουμε ότι, για παράδειγμα, η Ισπανία έχει ανάγκη γιατρικού προσωπικού. Γι' αυτό πρέπει να υπάρχουν εξειδικευμένοι γιατροί. Επίσης, να βλέπουμε και ποιες είναι οι ικανότητες και τα προσόντα των προσφύγων και των μεταναστών και να υπάρξει μια βάση δεδομένων η οποία να είναι ευρέως προσιτή. Η χρηματοδότηση χρειάζεται και για το Ευρωπαϊκό Ταμείο. Η Eurest θα κάνει διαχείριση και προσαρμογή ε, στα ευρωπαϊκά πρότυπα. Ο Υπουργό Απασχόληση θα είναι υπεύθυνο για να παράσχει τα στοιχεία τη χώρα του, ώστε να γνωρίζουμε ποιε είναι οι ανάγκε απασχόληση στου διάφορου τομεί. Αυτή η βάση δεδομένων έχει σαν στόχο τους μετανάστες και τους πρόσφυγες. Αλλά ε, θα πρέπει να, επίσης να προορίζεται και για τους άνεργους νέους. Θα πρέπει να γνωρίζουν ποιες είναι οι ευκαιρίες που προσφέρονται. Ε, πρέπει να υπάρχει μεγάλη διαφάνεια και να υπάρχει στρατηγική κατανομή ε, των μεταναστών. Υπάρχουν πολλά προσόντα σε όλη την Ευρώπη. Πρέπει λοιπόν όλοι μαζί να καταλάβουμε ποια είναι η αγορά εργασία για να αντιμετωπιστούν οι οικονομικές δυσκολίες. Επίσης μπορούμε να εντοπίσουμε ε, είναι, ποια είναι τα προσόντα και να καλύψουμε τα κενά ε, απασχόληση που υπάρχουν στις χώρες μας. Now I give the floor to our first MEP speaker. Δίνω τώρα ε, το λόγο στον πρώτο Ευρωβουλευτή ομιλητή, τον Τόμα Μάν, για δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ. Οι κατευθυντήριες γραμμές για τους νέους. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να πούμε ότι πρέπει να δώσουμε τη δυνατότητα σε όλους να δουν πραγματικά τι θέλουν να κάνουν. Είναι πολύ σημαντικό να ακουστούν λογικές προτάσεις, να δημιουργήσουμε προϋποθέσεις, να είναι γνωστοί οι κανόνες και βεβαίως κάθε φορά να γνωρίζουμε τις αξίες για την κάθε χώρα. Είναι επίσης πολύ σημαντική η πρακτική άσκηση, η εκπαίδευση, ναι, και πολλοί αυτό το έχουν πάρει από τις χώρες τους, από την οικογένειά τους, αλλά Κάναμε διάφορα πειράματα με νέους που προερχόταν από πολλές διαφορετικές ε, χώρες, πώς μπορούν να συνεργαστούν και να ζήσουν μαζί. Ποια είναι η δική σας ε, εμπειρία με νέους σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, παραδείγματο χάρη, είστε καλοδεχούμενοι, οι άλλοι που σας υποδέχονται εκεί, σας υποδέχονται με θετικό τρόπο η πολυπολιτισμική συνεργασία έχει επιτυχία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που λέτε για την ταχύτητα της διαδικασίας αναγνώρισης των διπλωμάτων, αναγνώρισης της επαγγελματικής ε, εμπειρίας ε, και των ε, διπλωμάτων. Αλλά βεβαίως είναι πολύ σημαντική η εκπαίδευση και τα διπλώματα, αλλά ακόμα πιο σημαντική, και αυτό στη Γερμανία πραγματικά το αξιολογούμε πολύ θετικά είναι η κατάρτιση, η πρακτική κατάρτιση. Και επίσης είναι πολύ σημαντικό κάποιος να συνειδητοποιεί ότι αυτή η πρακτική άσκηση, αυτή η κατάρτιση θα είναι σημαντικό και όταν ξαναγυρίσει πίσω στη χώρα του. Ευχαριστώ. Brandon Ο Brandon Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ για τις προτάσεις που ακούσαμε από τους νέους. Θα πρέπει να συνεχίσουμε αυτό το διάλογο, τον ξεκινήσαμε πέρσι και νομίζω ότι αυτή η πρωτοβουλία εδώ, στον οίκο της Δημοκρατίας, είναι κάτι που πρέπει να συνεχιστεί. Σαν εισηγητής για την ενσωμάτωση των μεταναστών στην αγορά εργασίας, γιατί ήμουν ο εισηγητής για την έκθεση με αυτό το θέμα. Βεβαίως και με έχει απασχολήσει το θέμα της αναγνώρισης των δεξιοτήτων αλλά και των διπλωμάτων, καθώς και την απόκτηση νέων διπλωμάτων και νέων ε, δεξιοτήτων. Αυτό είναι μια πρωτοβουλία που στηρίζουμε απόλυτα σαν Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και σε κάθε περίπτωση θέλουμε να υπάρξει καλύτερη εναρμόνιση ε, και εξομάλυνση μεταξύ των εκπαιδευτικών συστημάτων και της επαγγελματικής κατάρτισης των διαφόρων κρατών μελών. Υπάρχουν πολλοί φορείς, ιδρύματα του ιδιωτικού και του δημόσιου φορέα στις χώρες μας και σίγουρα χρειάζεται προσπάθεια ε, για να υπάρξουν οι αντιστοιχίες. Κατά την άποψή μου, θα πρέπει επίσης να γίνει μεγάλη προσπάθεια και επένδυση στον τομέα της ενσωμάτωσης, της καταπολέμησης της ε, ξενοφοβίας. Δεν μπορούμε να ενσωματώσουμε ανθρώπους εάν, ακόμα και αν υπάρχει αναγνώριση των δεξιοτήτων, παρά μόνο εάν δώσουμε νέες ευκαιρίες σε νέους, για καλύτερη κατάρτιση και για συνεχή ε, εκμάθηση νέων δεξιοτήτων. Αυτό αφορά τους νέους, αλλά όχι μόνο τους νέους και συμφωνώ με αυτό που είπατε ότι στα κράτη-μέλη θα πρέπει να υπάρξει καλύτερη ενημέρωση και ανταλλαγή στοιχείων. Το ίδιο όμως θα έλεγα και για την ίδια τη χώρα μέσα στην οποία πολλές φορές δεν υπάρχει συντονισμός μεταξύ των περιφερειών. Χρειαζόμαστε λοιπόν συντονισμό σε θεσμικό επίπεδο για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε αυτούς τους στόχους. Πρέπει το ευρωπαϊκό επίπεδο, το εθνικό επίπεδο και το περιφερειακό επίπεδο να συνεργαστούν με τις ενώσεις και τους φορείς που προωθούν τα δικαιώματα των νέων. Ευχαριστώ πολύ. Οι νέοι εδώ μας θέτουν πολύ συγκεκριμένα ερωτήματα και προκλήσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και είναι σημαντικό, ενώ μιλάμε για τους μετανάστες, οι οποίοι μπαίνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και οι οποίοι αντιμετωπίζονται με τελείως διαφορετικό τρόπο από τα κράτη-μέλη, οι μετανάστες που την χάνουν τελείως διαφορετικής υποδοχής από τη μία χώρα στην άλλη. Εμείς στη Γερμανία τους παίρνουμε πολύ σοβαρά υπόψη, αλλά βεβαίως υπάρχουν άνθρωποι που έρχονται από τελείως διαφορετικά περιβάλλοντα, από τελείως διαφορετικούς πολιτισμούς, μιλούν διαφορετικές γλώσσες. Μας ρωτάνε λοιπόν πώς μπορούμε να ενσωματωθούμε στις χώρες σας και στις κοινωνίες σας στην Γερμανία έχουμε ένα γενικότερο πλαίσιο με κατευθυντήριες γραμμές για την ενσωμάτωση των μεταναστών. Εσείς σαν νέοι μπορείτε να μας τροποδοτήσετε με στοιχεία. Είστε στην πρώτη γραμμή της διαργασίας αυτής και πολλές φορές βλέπουμε οι νέοι σήμερα από την Ευρώπη να φεύγουν, να πηγαίνουν στον Καναδά, στην Αμερική, στην Αυστραλία και εκεί μπορεί να υπάρχουν κάποιες πολιτισμικές διαφορές, αλλά πολύ λιγότερες. Ένας Αφρικανός νέος, ο οποίος έρχεται στην Ευρώπη, πρέπει να ενσωματωθεί, να μάθει τον πολιτισμό μας, να μάθει τα ήθη και έθιμα και πολλές φορές και τη γλώσσα. Εμείς καλούμεθα να κάνουμε την προσπάθεια να κατανοήσουμε γιατί η αφρικανική κοινωνία, παραδείγματος χάρη, είναι διαφορετικά οργανωμένη. Τι σημαίνει δουλειά στην Αφρική. Στις δικές μας πόλεις λοιπόν και στις δικές μας χώρες στην Ευρώπη θα πρέπει να γίνει προσπάθεια για να υπάρξει επιτυχής ενσωμάτωση των μεταναστών. Ευχαριστώ. Ο τελευταίος ομιλητής είναι η Ρενάτε Βέμπερ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Και ευχαριστώ πολύ τους συμμετέχοντες από το ΆΙ και επίσης για την εισαγωγή σας. Οπωσδήποτε συζητήσαμε το θέμα ε, των προσφύγων και των μεταναστών εδώ και ένα χρόνο και περισσότερο και μάλιστα εντατικά. Βεβαίω δεν έχουμε βρει ακόμα λύση. Τουλάχιστον όμω αναζητούμε μια λύση. Και με ευχαρίστηση σας άκουσα, παρόλο ότι ζούμε σε ένα παράδοξο. Αφενός, πολλές κυβερνήσεις λένε ότι τον έρχονται περισσότεροι πρόσφυγες στην αγορά εργασίας θα εμποδίσουν την είσοδο των νέων, της νέας γενιάς στην αγορά εργασίας. Βεβαίω μιλάμε διαφορετική γλώσσα. Το μήνυμά σα είναι διαφορετικό από εκείνο που ακούμε από επίσημου κύκλου σε όλη την Ευρώπη. Γι' αυτό το πρόβλημα τελικά είναι πολιτικό. Θα πρέπει να λυθεί σε πολιτικό επίπεδο πρώτα. Νομίζω ότι μια σημαντική πτυχή του θέματος είναι η πολιτιστική διαφορά. Υπό την έννοια ότι μπορεί να υπάρχει μια τάση στην Ευρώπη να αντιμετωπίζονται όλοι οι πρόσφυγες ομοίως. Είναι όμως διαφορετικοί, προέρχονται από άλλες περιοχές του κόσμου και φέρουν μαζί τους διαφορετική κουλτούρα. Το σημαντικό είναι για μας στην Ευρώπη να το καταλάβουμε ότι υπάρχει αυτή η διαφορά Γι' αυτό πιστεύω ότι χρειάζεται μια προσέγγιση στη βάση για να ενσωματωθούν στις κοινωνίες μας. Από την άλλη πλευρά, βεβαίως, έχει μεγάλη σημασία και τι δεξιότητες μας φέρνουν. Θα ήταν λυπηρό να μην χρησιμοποιήσουμε άτομα που έχουν τα προσόντα, διότι εμείς θα υποφεληθούμε από αυτό. Το ερώτημά μου λοιπόν προς εσάς είναι το εξής. Πώς νομίζετε ότι μπορείτε να περάσετε το μήνυμά σας στις κυβερνήσεις σας να εξηγήσετε ότι είσαστε ανοιχτοί και έτοιμοι να συνεργαστείτε με τους πρόσφυγες προκειμένου να ενσωματωθούν μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα ερχόμαστε πάλι ε, στους δύο αρχικούς ομιλητές που θα απαντήσουν στα ερωτήματα και στις ιδέες. Σε ομιλείτε, Λεωνή, εσύ πρώτα απ' όλα να απαντήσω στις δύο πρώτες ερωτήσεις. Οι φίλοι μου, από ό,τι ξέρω, είναι ανοιχτή σε άλλους πολιτισμούς και κουλτούρες. Εξάλλου, κάνουμε και αντιστοιχείες σπουδές εμείς στον Βασίλειο, που σχετίζονται με άλλες κουλτούρες και πολιτισμούς και όλη η δουλειά που κάνω αυτή τη στιγμή και μελέτη έχει διεθνή χαρακτήρα. Νομίζω είναι καλό να έχουμε άμεση επικοινωνία με μετανάστες. Γιατί δεν συναντάμε και πολλούς στο Σέφιλντ όπου μένω. Πρέπει λοιπόν να κάνουμε μια προσπάθεια επικοινωνίας με τους μετανάστες, να τους πούμε ότι είναι ευπρόζεκτοι στον δικό μας πολιτισμό και στην δική μας κουλτούρα, ώστε να υπάρχει αμοιβαία κατανόηση και να το στείλουμε αυτό σαν μήνυμα στην κυβέρνηση ότι είναι ευπρόσδεκτη στην κοινωνία μας και στην αγορά εργασία μας. Δεν ξέρω αν αυτό απαντάει το ερώτημά σας. Ευχαριστώ. Η Μελίσσα. Ναι, εγώ να κάνω δύο σχόλια για αυτό που είπατε για τη σημασία του πολιτισμού. Σκεφτόμουν την πρόταση του Γιούρας να υπάρχει δηλαδή ένα σύστημα όπου θα έχουμε μια προτίμηση θέλετε ας πούμε να πάτε στη Γαλλία να δηλαδή, δει ο πρόσφυγας ή ο μετανάστης τι ανάγκες υπάρχουν όσον αφορά τις δεξιότητές τους στην Ευρώπη και αντίστοιχα να μετακινηθούν. Να επιλέξουν λοιπόν τις δεξιότητές τους όχι μόνο καθοδόν και ανάλογα με τι ανάγκε, αλλά και τον πολιτισμό τους, την κοινωνία στην οποία θα ενταχτούν. Και αν εσείς πάτε σε μια πλατφόρμα αναζήτησης και δείτε ότι ας πούμε δεν υπάρχει, ότι δεν υπάρχει ανάγκη για τις δεξιότητές σας, τότε πρέπει να έχετε εναλλακτικέ. Να δείτε, ας πούμε, τι ανάγκες υπάρχουν σε άλλες χώρες και ταυτόχρονα να μάθετε και κάποια πράγματα για τον πολιτισμό αυτής της χώρας. Γιατί είναι αλήθεια ότι καμιά φορά βλέπουμε να λείπει συντονισμό σε αυτά τα θέματα και πρέπει να δίνεται ένα κίνητρο μέσα από τις στατιστικές και τα στοιχεία για τη χώρα ώστε να μπορεί κανείς να τα κοιτάζει και να μπορεί να εντοπίζει ας πούμε ό,τι και να υπάρχουν στις δεξιότητες και να προσπαθεί να τα καλύψει ώστε να υπάρχει δηλαδή ένα μεγαλύτερο κίνητρο και να δείξουμε στην κυβέρνηση ακριβώς πώς αυτοί οι μετανάστες, αυτοί οι άνθρωποι ωφελούν τη χώρα. Και δεν είναι μόνο θέμα δεξιοτήτων για αγορά εργασία. Ευχαριστώ. Ναι, είναι ταχεία αυτή η συνεδρία, οπότε προχωράμε. Θα περάσουμε στο δεύτερο γύρο ιδεών για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων ως μέσο αντιμετώπισης της ανεργίας των νέων. Λόρες Νόεν πρώτα για αυτό το θέμα. Δύο λεπτά. Αγαπητά μέλη του Κοινοβουλίου, αγαπητοί επισκέπτες, αγαπητοί θεατές online. Σήμερα βλέπουμε να λείπουν ψηφιακές δεξιότητες. Προτείνω λοιπόν να κάνουμε ένα καλοκαιρινό πανεπιστήμιο ψηφιακών δεξιοτήτων για τους νέους, ώστε να είναι ελκυστικοί στην αγορά εργασίας. Όσοι είναι άνεργοι θα πάρουν πρόσκληση για αυτό το καλοκαιρινό πανεπιστήμιο τεσσάρων εβδομάδων, ώστε μετά αυτή η εμπειρία να χρησιμοποιηθεί σε επιχειρήσεις και να γίνεται μάλιστα και δύο φορές ετησίως. Θα διδάσκονται προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών, λογισμικό και ανάλογα με αυτή την εξειδίκευση οι νέοι θα είναι σε θέση να επιλέξουν ένα κλάδο της βιομηχανίας, δηλαδή επιμελητία, παραγωγή κτλ. και αντίστοιχα να αποκτήσουν δεξιότητες λογισμικού. Βέβαια, θα υπάρχουν και τάξεις λογισμικού που θα διδάσκουν τα βασικά. Πάντω όλε οι τάξεις, αντίθετα με τις ε, τάξεις στο Πανεπιστήμιο, θα είναι διαδραστικές και θα περιέχουν και στοιχεία αυτοδιδασκαλίας. Θα πρέπει λοιπόν μαζί με τη μηχανία και τα πανεπιστήμια να διοργανώσουμε αυτά τα μαθήματα διατομιακά και κοντά σε επιχειρήσεις, κυρίως κοντά σε τοπικές επιχειρήσεις. Η χρηματοδότηση αυτών των μαθημάτων θα γίνεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα είναι δωρεάν για τους συμμετέχοντες. Για να βρούμε λοιπόν ένα βιώσιμο μοντέλο, 3-4-5 πανεπιστήμια θα μπορούσαν να ξεκινήσουν στην Ευρώπη αυτό το εγχείρημα, μαζί με κάποιες επιχειρήσεις, ώστε να μπορέσουμε να βελτιώσουμε αυτά τα μαθήματα και να προσελκύσουμε Νέου ώστε να αποκτήσουν αυτέ τι ψηφιακέ δεξιότητε. Ευχαριστώ πολύ. Thank you. And, uh, Ευχαριστώ πολύ. Τώρα, Ελένη, προτείνω η Ευρωπαϊκή Ένωση να υθετήσει ένα πλαίσιο για να προτρύνει τους παρόχους παιδείας, ούτως ώστε η μάθηση να είναι ευρεία. Αυτό θα επιτρέψει στη νέα γενιά να αντιμετωπίσει τις πολλές αλλαγές που επέρχονται χρειάζονται τρεις βασικές δεξιότητες, ακαδημαϊκές, τεχνικές και ε, επικοινωνιακές δεξιότητες και ομαδική δουλειά. Η ανεργία των νέων είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε σήμερα. Το ένα είναι ότι δεν υπάρχει αρκετή σχέση ανάμεσα στα όσα μαθαίνουμε στο σχολείο και αυτά που απαιτούνται στην αγορά εργασίας. Σήμερα είναι απαραίτητη αυτή η διασύνδεση. Η αγορά εργασία χρειάζεται άτομα να ενσωματωθούν, να έχουν ε, κοινωνική ευρωστία, να είναι ευέλιστα. Για... Δεν πρέπει να υπάρχει αυτό το κενό ε, στις δεξιότητες. Θα πρέπει να εκπαιδεύονται σε πραγματικές καταστάσεις. Θα πρέπει να συνδυάζεται με χρηματικά κίνητρα ούτω ώστε στη διάρκεια των σπουδών του οι νέοι να κάνουν και μαθητεία. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Μπόρεσα να κάνω δύο μαθητείες και αυτή ήταν μία από τις πιο σημαντικές αποφάσεις που είχα λάβει, διότι είδα τι περιμένει από μένα ένας εργοδότης και αυτό είναι πολύ πιο σημαντικό πιστεύω από τις νομικές γνώσεις που είχα. Επίσης, είχα μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στις ικανότητές μου να καταλάβω και να διεκπαιρεώσω θέματα, πράγμα που δεν μπορούσε να γίνει στο Πανεπιστήμιο. Επίσης, για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων θα πρέπει να βασιστούμε στις δεξιότητες που μαθαίνουμε κατά την εκπαίδευση, αλλά να δώσουμε μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση στους νέους για να βρίσκουν πρακτικές λύσεις στα προβλήματα και να έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να βρουν μια δουλειά. Ευχαριστώ. Thank you. Ευχαριστώ. Ο πρώτος ευρωβουλευτής από το γύρο είναι ο Hans Becker. Δύο λεπτά. Ευχαριστώ για αυτές τις παρουσιάσεις, οι οποίες πραγματικά ε, δένουν με αυτό το οποίο θα σας αναφέρω, 50 ιδέες ε, για την Ευρώπη. Εδώ και χρόνια δουλεύει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για αυτές ε, τις προτάσεις και ιδέες. Ε, εσείς μας κάνατε δύο πολύ συγκεκριμένες προτάσεις, τις οποίες στηρίζω 100% και για το θέμα των ψηφιακών δεξιοτήτων, αλλά και η δεύτερη ιδέα Το θέμα μας είναι να γίνουμε άτομα τα οποία να προσαρμοζόμαστε στις ανάγκες της αγοράς εργασίας, να γίνουμε απασχολήσιμοι. Δηλαδή η κατάρτιση θα πρέπει να ακολουθεί πρότυπα και μοντέλα τα οποία ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες. Αυτό που να καταλάβουμε όλοι μας εδώ. Η Επιτροπή 100 φορές έχει εξετάσει το θέμα αυτό και εκατό φορές έχει κατανοήσει ότι το θέμα της αγοράς εργασίας και της πολιτικής στον τομέα αυτό δεν είναι καθαρά αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και σε κάθε περίπτωση πολύ απλές ιδέες όπως ε, οι μαθητείες που δεν ανταμείβονται θα πρέπει να απαγορευτούν, πολύ απλά, να απαγορεύονται. Δεν είναι δυνατόν να υπάρχει ένα σύστημα το οποίο να επιτρέπει στις επιχειρήσεις και τους εργοδότες να ε, μην είναι κοινωνικά δίκαιοι. Θα πρέπει να δίνονται εγγύσεις στους νέους, να δούμε αν το υπάρχον σύστημα είναι επιτυχές, αποτελεσματικό και αυτό είναι κάτι που βέβαια Πολλές φορές δεν το κάνουμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοπούλιο, αλλά αυτή τη φορά θα ήθελα να συγχαρώ την Επιτροπή για αυτά που κάνει για το θέμα των soft power. Ευχαριστώ. Ο επόμενος Ευρωβουλευτής. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ για τις παρεμβάσεις και καλωσορίσατε όλοι και όλες. Εδώ συζητούμε με εσάς τους νέους αυτό το θέμα γιατί επειδή έχουμε μια Ευρώπη με 25 εκατομμύρια ανέργους και 7 εκατομμύρια άνεργους νέους. Πρέπει λοιπόν να αντιμετωπίσουμε την αιτία της ανεργίας και η αιτία είναι η έλλειψη ανάπτυξης. Εάν δούμε αντικειμενικά αυτό το θέμα, μπορούμε να πούμε τα τελευταία χρόνια οι ικανότητες των νέων στην Ευρώπη παρουσιάζουν αύξηση. Λοιπόν, ε, εκείνο το οποίο κατηγορούμε δεν είναι το νέο, όχι για, τον, ε, ε, για την έλλειψη ικανότητας, αλλά την έλλειψη εμπειρίας. Και εδώ βρίσκεται το πρόβλημα. Και παρακολούθησα με μεγάλη προσοχή και ενδιαφέρον αυτά τα οποία ελέγχθησαν ανάμεσα στη συσχέτιση μεταξύ του κόσμου της εκπαίδευσης και του κόσμου της εργασίας. Χρειάζεται μεγάλη συνεργασία μεταξύ των δύο προκειμένου η εκπαίδευση να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των επιχειρήσεων. Και Τη αγορά εργασία. Γι' αυτό πρέπει να διαχειριστούμε σωστά ε, τις ικανότητες των νέων. Αυτό βεβαίω έχει σχέση με την ευρωπαϊκή πύλη που πρότεινε η Μελίσσα. Είναι η ίδια ιδέα. Δηλαδή οι επιχειρήσει πρέπει να μα πούν εκ των προτέρων ποιε θα είναι οι ανάγκε του σε 5, 6, 7 χρόνια ώστε εμεί να προλάβουμε. Και το ανησυχητικό, δραματικό είναι για μας ε, τους ε, γονείς και εγώ έχω δύο παιδιά που ψάχνουν δουλειά και δεν είναι ότι δεν έχουν προσόντα αλλά δεν έχουν πείρα. Λοιπόν οι επιχειρήσεις συχνά θεωρούν ότι είναι κίνδυνο να προσλάβουν ένα νέο, επειδή δεν είναι λειτουργικός άμεσα. Και εδώ θα πρέπει η Ευρώπη να χρησιμοποιήσει κίνητρα, διότι μερικές φορές ε, η μαθητεία γίνεται σε επιχειρήσεις, αλλά δεν είναι πάνω το δυνατή. Χρειάζονται κίνητρα λοιπόν, ώστε οι επιχειρήσεις να δεχτούν να προσλάβουν ένα νέο, ώστε για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα, έξι μήνες, ένα χρόνο, να, να μάθει τη δουλειά και να ε, να έχει κοντά του έναν αρχαιότερο που θα του, μάθει, τη δουλειά. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Um, Ευχαριστώ. Δεν βλέπω την Τόνια Κονσάλες εδώ. Οπότε, τον Ιρανικά, επόμενη ομιλήτρια. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εγώ να σας καλωσορίσω θερμά όλους και όλες. Θαυμάσια στιγμή. Θυμάμαι μετά την τελευταία μας συνάντηση που ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα έμεινα με τις καλύτερες εντυπώσεις και δεν είμαι και τόσο μακριά ηλικιακά από σας. Χαίρομαι λοιπόν που έχουμε τόσους νέους εδώ σήμερα και που συζητάμε. Μετά από αυτά που υπόθηκα να σας πω κι εγώ ότι με ενδιαφέρει πολύ η πρόταση για το Θερμινό Πανεπιστήμιο Ψηφιακών Δεξιοτήτων και θα μπορούσαμε να το προτείνουμε πιλωτικά ως πρόγραμμα για του χρόνου ώστε να εφαρμόσουμε αυτά τα μοντέλα σε διάφορα πανεπιστήμια όπως πρότεινες. Και μου αρέσει αυτή η ιδέα επειδή ακριβώς ενισχύει τους νέους. Και αυτά ακριβώς ήθελα να πω και εγώ και θα ήθελα τα σχόλιά σας. Ίσως να διαφωνήσω για το ότι οι δεξιότητες και η εκπαίδευση θα πρέπει να αφορμούν την αποσχολησιμότητα των νέων. Νομίζω ότι αυτά τα δύο θα πρέπει να είναι κάτι παραπάνω. Δηλαδή θα πρέπει να μιλάμε για την προσωπική εξέλιξη των ατόμων, των νέων ατόμων, την δημιουργία ελεύθερου χώρου στη ζωή μας, την ανάπτυξη της προσωπικότητας. Παρόλο λοιπόν που υπάρχουν αποκλήσει όσον αφορά τι δεξιότητε, να μην το ξεχνάμε αυτό, γιατί αυτοί ακριβώς είναι οι χώροι που οι νέοι δεν μαθαίνουν μόνο να είναι τμήμα τη αγορά εργασία, αλλά μαθαίνουν και δεξιότητε δημοκρατικέ και πολιτική αγωγή. Αυτό είναι σημαντικό για την κοινωνία. Το επόμενο που θα ήθελα να αναφέρω, διαφωνώντας σε σχέση με αυτά που είπατε, είναι το εξής. Μιλάμε για έλλειψη δεξιοτήτων. Αν δείτε την πραγματικότητα, νομίζω ότι είμαστε οι πιο εξοπλισμένοι με προσόντα γενιά. Οπότε περιμένουμε τις δημόσιες επενδύσεις για δημιουργία θέσεων εργασίας, για την απασχόληση αυτών των νέων. Θα θέλαμε λοιπόν η Ένωση να κάνει κάποια πράγματα. Εσείς τι προσδοκίες έχετε γι' αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ε, παραρχόμαστε τώρα για ένα λεπτό στους ηγητές μας. Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ιδέες της δικές σας και τα σχόλιά σας. Συμφωνώ. για το ότι λείπει η προσωπική εξέλιξη. Στη Γερμανία οι σπουδές είναι θεωρητικές και οι πρακτικές δεξιότητες λείπουν. Οπότε η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να συμβάλλει, έστω και με ένα μικρό ποσοστό, 5-10% στην προσωπική εξέλιξη. Εγώ σπούδασα και στο Παρίσι. Οι σπουδές ήταν τελείως διαφορετικές, διατομιακές, διακλαδικές. Δεν είχαν στόχευση μόνο σε ένα μάθημα, και είχαν διαφορετικό προσανατολισμό. Αλλά βλέπουμε και την επικράτηση της θεωρίας. Και έχουμε πάντως θετικά παραδείγματα, τα οποία έχουν εφαρμοστεί και στη Γερμανία, τα οποία θα μπορούσαν να έχουν θετικό αντίκτυπο στην Ευρώπη. Τώρα για την απόκληση που λέγαμε στις δεξιότητε δεν είναι τόσο η λήψη, όσο διαφορά ταυτότητας των δεξιοτήτων. Εμείς θα πρέπει λοιπόν να ρωτήσουμε τους εργοδότες τι προσδοκούν, τι αναμένουν από τους φοιτητέ στο τέλος των σπουδών τους. Λεωνί, έχεις ένα λεπτό κι εσύ. Να απαντήσω σε κάποια από τα σημεία. Κύριε Μπέκερ, συμφωνώ απολύτως με αυτό που είπατε. Πρέπει να απαγορευτούν οι δωρεάν και οι ε, άμυστες μαθητείες. Γιατί βλέπουμε ότι τελικά κάποιος με πτυχία ουσιαστικά τελειώνει τις σπουδέ του μετά από τρία χρόνια και πρέπει να συνεχίσει και ξέρουμε ότι οι σπουδέ ε, κοστίζουν. Θα συμφωνήσω επίσης ότι είναι πολύ σημαντική η προσωπική εξέλιξη, η ανάπτυξη των προσωπικών ε, δεξιοτήτων και ικανοτήτων, πολύ περισσότερο από την εκπαίδευση αυτή καθεαυτή και την ε, δυνατότητα να ενσωματωθεί κανείς στην ε, αγορά εργασίας. Πολλές φορές τα προσόντα που διαθέτουμε, αυτά δηλαδή που αποκτούμε κατά τη διάρκεια των σπουδών μας και της ζωής μας, είναι προσόντα τα οποία προέρχονται εκτός των σπουδών. Δεν ξέρουμε πώς να τα χρησιμοποιήσουμε. Δεν ξέρουμε, ε, παραδείγματο χάρη, τι ακριβώς διαθέτουμε και πώς να τα αξιοποιήσουμε. Εγώ, ας πούμε, σπουδάζω νομικά. Και όταν με ρώτησαν σε μια συνέντευξη αν έχω εμπειρία σε θέματα marketing, η απάντησή μου είναι όχι και πώς θα μπορούσα να αποκτήσω εκτός των σπουδών μου και εκτός του πτυχίου μου. Ε, είναι λοιπόν πολλές φορές δύσκολο κανείς κάποια πράγματα που ενδεχομένως τα έχει και τα ξέρει να τα παρουσιάσει και να ε, τα χρησιμοποιήσει. Πρόεδρος, περνάμε στο τρίτο θέμα που είναι η νέα επιχειρηματικότητα και οι startups. Η Μελίσσα έχει το λόγο για δύο λεπτά. Πώς μπορεί κάποιος να μιλήσει για τους νέους επιχειρηματίες, να τους βοηθήσει. Προτείνουμε λοιπόν μία θηρίδα, one-stop shop, για να δίνονται πληροφορίες σε όλους αυτούς που θέλουν να δημιουργήσουν μία μικρή επιχείρηση, μία startup. Χρειάζονται πληροφορίες ε, που να βοηθούν αυτούς που δεν μιλούν τη γλώσσα της χώρας να μπορούν να κάνουν τις διοικητικές διαδικασίες, θα πρέπει επίσης να συγκεντρώνονται όλα τα προσωπικά δεδομένα, να δίνονται πληροφορίες για τον τομέα, για τον κλάδο και βεβαίως πληροφορίες όσον αφορά την χρηματοδότηση των επιχειρήσεων με έναν απλοποιημένο τρόπο και να δίνονται οι δυνατότητες ε, στους επιχειρηματίες, στους νέους επιχειρηματίες να δραστηριοποιηθούν χωρίς υπερβολικό βάρος διοικητικό και οικονομικό για τους πρώτους έξι μήνες ή χρόνο της ίδρυσης της επιχείρησής τους. Είναι η μεγαλύτερη πρόκληση που πρέπει να ε, αντιμετωπίσουμε και είναι πολύ σημαντικό να δούμε αν υπάρχει πάντα αντιστοιχεία μεταξύ του τομέα και του επιχειρηματία. Νέοι επιχειρηματίες όπως εγώ θέλουν να καταλαβαίνουν πώς λειτουργεί ε, το δίκτυο, πώς μπορούν να συλλέξουν τις απαραίτητες πληροφορίες και βεβαίως να εξοικονομήσει χρόνο για ό,τι αφορά τις διοικητικές διαδικασίες και την γραφειοκρατία. Αυτό βεβαίως ε, μας οδηγεί στη διαπίστωση ότι η κατάσταση είναι τελείως διαφορετική από τη μια χώρα στην άλλη. Η, τα δίκτυα υπάρχουν και λειτουργούν λίγο πολύ ικανοποιητικά στα κράτη-μέλη. Η καλύτερη χρησιμοποίηση της χρηματοδότησης είναι επίσης μία από τις εγγύσεις αποτελεσματικότητας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Επόμενο, επόμενο θέμα και ο Έχουμε το σχέδιο απασχόληση 2020. Θα ήθελα λοιπόν να, ζητήσουμε να δημιουργήσουμε μια ευρωπαϊκή πλατφόρμα για τις startups που θα μπορούσε να εφαρμοστεί τοπικά στα πανεπιστήμια ώστε να μπορούν να συναντιούνται οι υποψήφοι και να επιχειρούν. Πώς θα δουλεύει. θα είναι online αυτή η πλατφόρμα και θα μπορεί ο καθένας να δημιουργεί, να δημοσιεύει ιδέες επιχειρηματικές εκεί, ώστε και οι υπόλοιποι να μπορούν να δουν τις ιδέες αυτές, ανάλογα με το περιεχόμενο και το αντικείμενο. Να υπάρχει συγκεκριμένο αριθμό ατόμων που θα συμμετέχουν σε αυτή την προσπάθεια και να συνοδεύεται η προσπάθειά τους από κονδύλια. θα διατίθεται χώρος εργασίας στους επιχειρούντες από τα πανεπιστήμια και επιπλέον οι παλαιοί επιχειρηματίες μπορούν να λειτουργήσουν ως μέντορες για αυτούς τους νέους επιχειρηματίες των startups. Επίσης, εκτός από αυτή την πλατφόρμα, προτείνω να δημιουργηθεί μια πανευρωπαϊκή πλατφόρμα για τις startups για ανταλλαγή εμπειριών και πληροφοριών. Αφού λοιπόν δημιουργηθούν, μπορούν να εφαρμοστούν σε ξένες αγορές, ώστε να έχουμε γνώσεις και πληροφορίες για αντίστοιχους επιχειρηματίες σε άλλες χώρες και σε άλλες υπήρους. Μπορεί να γίνει μετά ανταλλαγή εκτός από πληροφοριών και στοιχείων και εργαζομένων. Θα πρέπει επίσης να επιλέγονται οι τρεις πιο υποσχόμενες επιχειρήσεις της πλατφόρμας και βεβαίως θα μπορούσαν να αντέχονται και βραβεία και έπαθλα. Αυτά θα αποτελέσουν νομίζω πολύ καλό παράδειγμα για τους νέους, ιδιαίτερα στην Ευρώπη, ώστε να ε, λάβουν κάποια κίνητρα να επιχειρούν περισσότερο. Ευχαριστώ πολύ. Thank you, Lawrence. Now... Ευχαριστώ πολύ, Lawrence. Τώρα ερχόμαστε στους δύο ευρωβουλευτές. Πρώτα Σέντσουλ για δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους νέους για τη συμμετοχή τους. Οι δηλώσεις τους είναι πολύ ενδιαφέρουσε, πρόκειται για ενδιαφέρουσε και ωραίες προτάσεις που καταδεικνύουν ότι σκεφτήκατε πολύ το θέμα Προσωπικά αυτό το θέμα των νεοφιών επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών με ενδιαφέρει πολύ, διότι πρόκειται για ένα σημαντικό στοιχείο για την Ευρώπη. Συζητήσαμε πολλά θέματα και ο τρόπος τον οποίο παρουσιάσατε την κατάσταση ήταν πολύ ενδιαφέρουσα. Μιλήσατε για πλατφόρμες online, ανταλλαγή καλών πρακτικών. Αυτά ακριβώς ζητούμε στην έκθεσή μας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιθυμούμε όλοι να συζητούν μεταξύ τους και να ανταλλάσσουν ιδέες. Αυτά τα δίκτυα λοιπόν είναι πολύ χρήσιμα. Πολλές νεοφυείς επιχειρήσεις αποθαρρύνονται από τη γραφειοκρατία που τους εμποδίζει να αναπτυχθούν. Ένα άλλο σημαντικό είναι ότι πρέπει να δημιουργήσουμε ένα λόμπι για τις νεοφυείς επιχειρήσεις είναι σημαντικό να πούμε ότι, ε, να τους πούμε ότι μπορεί να αποτύχετε, αλλά να ξεκινήσετε από το μηδέν. Όταν αποτυγχάνει κανείς, δεν είναι πραγματική αποτυχία, δεν είσαι χαμένος, επειδή αποκομίζεις εμπειρίες. Στη Γερμανία, τη χώρα μου, οι περισσότεροι νέοι προτιμούν να γίνουν υπάλληλοι, ε, δημόσιοι υπάλληλοι, διότι έχουν ασφάλεια για όλη τη ζωή. Αλλά θα έπρεπε το αντίθετο ε, να συμβαίνει. Οι νέοι πρέπει να έχουν το θάρρο να αναπτύξουν δραστηριότητες και πρωτοβουλίε και γι' αυτό πρέπει να του βοηθήσουμε. Με δύο λόγια, η χρηματοδότηση Μπορεί να υπάρξει, υπάρχουν χρήματα και πολλοί είναι διατεθειμένοι να χρηματοδοτήσουν τους νέους, ε, την πρωτοβουλία των νέων. Ο κ. Πέκερ είχε μια ενδιαφέρουσα ιδέα. Θα πρέπει να απαγορεύονται σε Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να γίνονται στάζ που δεν αμείβονται. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Μίλαν Παβό, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για τις ωραίες ιδέες που διατυπώσατε για Όλες οι προτάσεις σας είναι πολύ ενδιαφέρουσες και πιστεύουμε ότι θα κατορθώσουμε να τις αξιοποιήσουμε στο μέλλον. Θα πρέπει οι Ευρωπαίοι επιχειρηματίες να είναι οι παγκόσμιοι ηγέτες. Είναι κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Δεν πρέπει να είμαστε καταναλωτές προϊόντων που παράγουν οι άλλοι. Αν θέλουμε λοιπόν να γίνουμε ηγέτες σε αυτό το χώρο, θα πρέπει να ενθαρρύνουμε τη νέα γενεά να ξεκινήσει τις δικές επιχειρήσεις να γίνουν νέοι επιχειρηματίες, το οποίο σημαίνει ότι και επενδύτε και τραπεζίτες θα πρέπει να δώσουν πιστώσεις στους νέους, ακόμα και αν οι νέοι αποτύχουν. Ακόμα και αν γνωρίσουν μία ή δύο αποτυχίες. Υπάρχουν πρότυπα τα οποία μπορούμε να τους δείξουμε το Τελαβίδ και Silicon Valley, αλλά πιστεύω ότι δεν πρέπει να επαναλάβουμε τα υπάρχοντα μοντέλα. Θα πρέπει να εστιάσουμε περισσότερο στην ε, αναβάθμιση των ε, προσόντων και των δεξιοτήτων των νέων και να τους προσφέρουμε χρηματοδότηση. Μιλήσατε για ψηφιακές δεξιότητες. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και θα πρέπει να τους παροτρύνουμε να ακολουθήσουν αυτή την κατεύθυνση. Εγώ είμαι μηχανικός και ξέρω πολύ καλά το θέμα αυτό είναι αναγκαίο να, αναβαθμιστούν οι ικανότητες, οι ψηφιακές ικανότητες των νέων. Επίσης πρέπει να αντιληφθούμε ότι οι νεοφύης επιχειρήσεις έχουν άλλο επιχειρησιακό μοντέλο από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Πρέπει να το δούμε αυτό, να το λάβουμε υπόψη και να το περιλάβουμε στο νομοθετικό μας πλαίσιο, δηλαδή να προβλέψουμε τις ανάγκες των νεοφυών. Δεν έχω άλλο χρόνο, αλλά θα ήθελα τέλος εξίσου σημαντικό να προσθέσω, πρέπει να, τους, να παροτρύνουμε συνεργασία μεταξύ νοφιών επιχειρήσεων και πανεπιστημίων, ώστε να γίνουν τα φυτόρια όπου θα απελευθερωθεί η καινοτόμως δραστηριότητά τους. Ευχαριστώ πολύ. Thank you. And Και ο τελευταίος, η τελευταία ομιλήτρια είναι η Λόρα Άκλη. Δύο λεπτά. Καλημέρα σε όλους. Σας ευχαριστώ για τις εισηγήσεις σας. Επειδή προσφέρετε ένα φως πιο εξειδικευμένο σε σχέση με τις ανάγκες σας. Ιδιαίτερα με τον τρόπο που ερμηνεύετε την πραγματικότητα. Χρειαζόμαστε λοιπόν τη νέα φρέσκια ματιά σας για θέματα όπως ας πούμε η startup. Εγώ συχνά ήρθα σε επαφή με νέους και με το επιχειρηματικό τους πνεύμα που συχνά όμως αντιμετωπίζουν μια πραγματικότητα που κάνει δύσκολο το να γίνουν υλοποιήσιμες κάποιες ιδέες. Οι startups σήμερα αντιμετωπίζουν διάφορα προβλήματα επειδή η πρόσβαση στις πιστώσεις είναι ιδιαίτερα δυσχερής όπως επίσης και η γραφειοκρατία που αντιμετωπίζουν οι νέοι επιχειρηματίες είναι έντονη και οι δυσκολίες αυτές οι γραφειοκρατικές τους αποτρέπουν από το να υλοποιήσουν τα σχέδιά τους. Οι Μιλάμε και για διόδους χρηματοδότησης που είναι διαφορετικές από αυτές που προτείνατε εσείς, όπως τα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Τραπέζας Επενδύσεων. Οι νέοι που θέλουν να ανοίξουν startup πάνε στο business angel και στο crowdfunding. Και σωστά υποβάλατε τα αιτήματα που ακούσαμε προηγουμένως. Θα ήθελα εδώ λοιπόν να το τονίσω αυτό, όπως επίσης και το ότι πολύ συχνά ακούσαμε και είδαμε μεγάλες ιδέες που αναπτύχθηκαν από νέους, που δυστυχώς στη συνέχεια απολύθηκαν σε πολυεθνικές. Θα έπρεπε λοιπόν να δώσουμε περισσότερη έμφαση στην συνέχεια. Αν η ιδέα πρόκειται από ένα νέο, θα ήθελα να την διατηρήσει και όχι να την πωλήσει ο νέος αυτός σε άλλους. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Για ένα λεπτό οι δύο ομιλητές μας, οι δύο εισηγητές μας για αυτό το θέμα, η Μελίσσα πρώτα. Για το τελευταίο που είπατε, για την πώληση των startups, αυτό που είναι σημαντικό η χορηγοί και μέντορες αυτοί δηλαδή που βοηθούν τους νέους είναι σημαντικό να είναι από πολύ μεγάλες επιχειρήσεις ιδιαίτερα αν δείχνουν εμπιστοσύνη και πιστεύουν τους νέους και τις ιδέες τους γιατί είδαμε περιπτώσεις χρηματοδότηση επιχειρήσεων που οδήγησαν στην έξοδο τους νέους που δημιούργησαν τις startups. Τι άλλο, είχα εδώ ένα λεπτάκι. Α, ναι. Δεν νομίζω ότι είναι η ίδια γραφειοκρατία αυτή, κάθε αυτή που είναι σημαντικό ζήτημα. Πιστεύω ότι θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα να κατανοήσουμε ότι φοβίζει καμιά φορά η διαδικασία δημιουργίας startups αλλά θα πρέπει ακριβώ να κατανοήσουμε ότι αυτή η δημιουργία τη επιχειρηματικότητα αφορά όλου μα. Δεν είναι για λίγου και εκλεκτού. Ναι, και εγώ για τι δεξιότητε να πω έχουμε ένα μεγάλο οργανισμό στην Γερμανία που βοηθάει ακριβώ τις δεξιότητε, είδα ένα πρόσωπό τους χθε και μα είπε ότι ακριβώ κάνουν σεμινάρια, κατάρτιση, εκπαίδευση κτλ. Είναι λοιπόν σημαντικό να υπάρχει δυνατότητα έναρξη αυτών των επιχειρήσεων, αλλά θα πρέπει να συνοδεύονται αυτέ τι δραστηριότητε από μαθήματα καινοτομία, ενδεχομένω πανεπιστημιακό επίπεδο, ώστε να βοηθηθούν αυτοί οι άνθρωποι. Επίση, με ενδιαφέρει αυτή η επιχειρηματικότητα, αφού είδα ότι πολλέ startups ξεκίνησαν από άτομα που ήταν συμφιλητέ μου είναι καλό λοιπόν να ξεκινούν αυτές τι προσπάθειε για startups, αλλά ήδη να συνοδεύονται από εκπαιδευτικά προγράμματα ήδη από τα πανεπιστήμια και σε μία επιμόρφωση επιχειρηματικά, αντί να γίνονται αυτά στο τέλος. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, Λαϊκή Πρόεδρος. Θα ζητήσω από του καημένου τους να δείξουν υπομονή πέντε λεπτάκια. Είναι σημαντικό να ακούσουμε την εκπρόσωπο της Κομισιόν, την Γενική Διευθύντρια της Κομισιόν, η Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης. Σας καλωσορίζω και σας το λόγο αμέσως για λίγα λεπτά. Θα προσπαθήσω να είμαι όσο δυνατόν ε, συντομότερος. Πρώτα απ' όλα ευχαριστώ πολύ για τις νέες ιδέες που προσφέρατε δεν συμβαίνει συχνά να ακούμε νέες ιδέες και τις χαιρετίζω, κυρίως τη στιγμή που χρειάζεται νέες προσεγγίσεις, νέες μεθόδους και νέες ιδέες η Ευρώπη. Ας ξεκινήσω με τη μετανάστευση. Πρώτα απ' όλα θεωρώ καθησυχαστικό να ακούω πόσο οι νέοι υποστηρίζουν τη μετανάστευση. Αυτό είναι θετικό, διότι εκείνοι που είναι περισσότερο εκτεθειμένοι στην παγκοσμιοποίηση είναι οι νέοι. Το γεγονός ότι αντιλαμβάνονται τα θετικά στοιχεία της μετανάστευσης είναι κάτι το σημαντικό. Επίσης, θα ήθελα να σας πω ότι για την Ευρωπαϊκή Ένωση εμείς βασιζόμαστε ε, στην ποικιλομορφία, στη διαφορετικότητα. Πρέπει να καταλάβουμε λοιπόν πώς να αναγνωρίζουμε τη διαφορετικότητα και να την ενσωματώνουμε. Τώρα, όσον αφορά η ενσωμάτωση, την ενσωμάτωση στην αγορά εργασία, θα να σα πω το εξή. Τώρα υπάρχει αυτή η μεταναστευτική ροή που είναι δύσκολο να αντιμετωπιστεί για ορισμένα κράτη-μέλη Το σημαντικό εδώ είναι να αντιμετωπίσουμε ανεπίσημα αυτό το θέμα Πρακτικά όμως, όσον αφορά τις δεξιότητες, δεν μπορείτε να αναμένετε ότι θα χρησιμοποιείτε αυτή η τυπική διαδικασία. Ε, το σημαντικό είναι να βρούμε ένα σύστημα όπου μπορούμε να δοκιμάσουμε τις δεξιότητες ε, και τις αρμοδιότητες, τις ικανότητες εκείνων που έρχονται και να βρούμε μια γρήγορη διαδικασία για να επισημάνουμε τις ικανότητές τους. Πρέπει λοιπόν να είμαστε ευέλικτοι, πρακτικοί και να εξασφαλίσουμε ότι εκείνοι που φθάνουν έχουν τη δυνατότητα να ενταχθούν στην αγορά εργασία το ταχύτερο δυνατόν. Όσον αφορά τις δεξιότητες, συμφωνώ ότι οι ψηφιακές δεξιότητες είναι σημαντικές. Για μένα η ο αλφαβητισμός και οι γνώσεις των υπολογιστών είναι πολύ σημαντικές. Έχουμε 17 εκατομμύρια άτομα τα οποία ε, σημαίνουν το μέγεθος της χώρας μας. Είναι πάρα πολλοί αυτοί οι άνθρωποι. Να σκεφτείτε ότι παρουσιάζουν ένα μεγάλο πρόβλημα, διότι αν θέλουν να ενταχθούν στην αγορά εργασίας, χωρίς να ξέρουν από κομπιούτερ, χωρίς να έχουν, ξέρουν γράμματα ε, και αριθμούς σωστά δηλαδή, είναι δύσκολο να βρουν δουλειά. Γι' αυτό ε, προτείνουμε εγγύηση δεξιοτήτων. Συμφωνώ μαζί σας ότι η λύση των προβλημάτων είναι κάτι το απαραίτητο για το μέλλον. Οι νέοι θα περάσουν από μια δουλειά στην άλλη στο μέλλον. Συνεπώς το ζητούμενο δεν είναι πώς να γίνει κανείς ξυλουργός. Το ζητούμενο είναι πώς να μπορεί να αλλάξει δουλειά από ξυλουργός ε, σε υδραυλικό ή σε τεχνικό κομπιούτερ. Τέλος, όσον αφορά τη σύνδεση ανάμεσα στην εκπαίδευση, στο εκπαιδευτικό σύστημα και τον εργοδότη. Στην Επιτροπή σκεφτήκαμε και το δουλεύουμε αυτό, πώς να υπάρξει, να ταιριάζουν οι, οι, οι εκπαιδευτικές ικανότητες με τη δουλειά αλλά πρέπει να το δούμε και από τη σκοπιά των νέων, διότι οι νέοι θα πρέπει να κάνουν τη διασύνδεση ανάμεσα στις γνώσεις τους, στην εκπαίδευσή τους, στην παιδεία τους και στην εργασία τους σε μια εταιρεία. Νομίζω ότι ένας από τους νέους είπε ότι το να φτάσει κανείς σε μια εταιρεία, τότε την έκανε να καταλάβει τι, τι ζητάει ο εργοδότης. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Γι' αυτό κοιτάμε πώς θα εξασφαλίσουμε κινητικότητα για τους μαθητευόμενους και ποιο θα είναι το σχέδιο στο μέλλον, η δομή στο μέλλον ε, που η κατάλληλη για νέους επαγγελματίες, διότι πιστεύουμε ότι αυτή η εμπειρία είναι αυτό το οποίο χρειάζεται. Τέλος, για την επιχειρηματικότητα. Εντυπωσιάστηκα πριν από δύο χρόνια από μια μελέτη που δημοσιεύτηκε και έδειχνε ότι οι απόφοιτοι πανεπιστημίου, μόνο το 30% εξ αυτών σκέφτονται να γίνουν επιχειρηματίες. Εάν γίνει η ίδια μελέτη στις ΗΠΑ, η στεντρική πλειοψηφία, το 70%, θέλουν να γίνουν ανεξάρτητοι επαγγελματίε, επιχειρηματίε δηλαδή. Αυτή είναι μια μεγάλη διαφορά και αυτό είναι το πρόβλημα. Η ιδέα των επιχειρησιακών δικτών είναι πολύ σημαντική, ήδη υπάρχει σε ορισμένα κρατημέλη, αλλά πρέπει να είναι κάτι το οποίο συστηματικά θα εφαρμόζεται σε όλα τα πανεπιστήμια. Και αυτό όχι μόνο για τις ε, νεοφύης επιχειρήσεις, αλλά και για τις άλλες. Διότι δηλαδή, το πρόβλημα της νεοφύης επιχειρήσεις είναι πώς θα γίνουν μια πραγματική επιχείρηση. Λοιπόν υπάρχει αυτή η απόκληση ανάμεσα σε την επιχείρηση και στη μικρομεσαία επιχείρηση. Τα πανεπιστήμια είναι σημαντικά, θα πρέπει να δούμε τις νοφείς επιχειρήσεις σε ένα ευρύτερο πλαίσιο. Γιατί για μένα αυτό δεν αφορά μόνο τα πανεπιστήμια. Αυτό το οποίο συζητάμε τώρα είναι οι μικροπιστώσεις, η δημιουργία ε, επιχειρήσεων, μικροεπιχειρήσεων, ένα μικρό εστιατόριο, ένα μικρό κομμωτήριο και ούτω καθεξής, να προωθηθούν όλες οι επιχειρησιακές δυνατότητες. Θα ήθελα να πω ότι μου αρέσει η ιδέα του one-stop shop, διότι πρόσφατα ήθελα να δω πώς μπορεί να γίνει κανείς αυτοαπασχολούμενος στη χώρα μου. Λοιπόν, ε, επισκέφθηκα ένα-δύο μια-δύο ιστοσελίδε και ε, όχι επειδή είμαι μεγάλη ηλικία, αλλά είδα αρνητικά, αν θέλετε, τη γραφειοκρατία που πρέπει κανείς ε, να περάσει όσον αφορά τα λογιστικά, την επιστροφή φόρων και ούτω καθεξής. Λοιπόν, η ιδέα του one-stop shop είναι πολύ σημαντική. Ένα σημείο όπου ένας δυνητικός επιχειρηματίας θα βρει όλα τα διοικητικά και θα λύσει όλα τα γραφειοκρατικά προβλήματα προτού ξεκινήσει την επιχείρησή του. Λυπούμε, λοιπόν, προσπάθησα να καλύψω όλα τα θέματα και τα κάλυψα με μεγάλη ταχύτητα, αλλά γνωρίζω ότι έχετε περιορισμό χρόνου. Ευχαριστώ που μου δώσατε το λόγο. Ευχαριστούμε. Έχουμε δυστυχώς ξεπεράσει το χρόνο μας. Ευχαριστώ τους τρεις ομιλητές, τους τρεις νέους που είναι σήμερα εδώ και τις εξαιρετικές προτάσεις τους. Ευχαριστώ και όλους τους άλλους για την υπομονή τους. Νομίζω πραγματικά ότι είναι μία από τις καλύτερες ακροάσεις που είχαμε εμείς σαν Επιτροπή Απασχόλησης και ελπίζω να κάνουμε κι άλλες τέτοιες ακροάσεις. Πραγματική έμπνευση για όλους μας. Εγώ ξεκίνησα πραγματικά την επιχείρησή μου στα 22 μου και χαίρομαι γιατί βλέπω ότι άλλοι νέοι επιθυμούν να κάνουν το ίδιο. Ό,τι μπορούμε να κάνουμε εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να στηρίξουμε τους νέους επιχειρηματίες θα το κάνουμε. Ευχαριστώ πολύ και σας καλώ όλους για ένα ποτήρι, για ένα ποτό έξω από την αίθουσα.